Ξεκινάμε αμέσως διότι έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον παλιό συνάδελφο και τον ευχαριστούμε που δέχθηκε την πρόσκλησή μας να μιλήσει για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρεις πολύ καλά το κοινοβούλιο, ξέρετε πολύ καλά το, το κοινοβούλιο σήμερα, σπίτι σας είστε, έχουμε πολλά ζητήματα. Ξέρετε πολύ καλά τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, όπως γνωρίζετε. Εμείς θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι στο κέντρο των πολιτικών συζητήσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είσαστε ένα επίτιμο μέλος το ποντινά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά τη, αυτό το καλωσόρισμα σας δίνω απευθείας τον λόγο και ευχαριστώ εκ νέου για την παρουσία σας εδώ. Ε, ε, Άρχεται η ηλεκτρονική διαδικασία για το Catch the Eye. Μετά τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού κ. Κάριντς. augsti godātais tajani kungs prezident juncker kungs Κύριε Πρόεδρε Ταγιάννη, κύριε Πρόεδρε και κύριοι φίλοι. Καταρχήν, ιδιαίτερα που σας μιλώ για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, το μέλλον της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για δέκα χρόνια περίπου, εργάστηκα, ήμουν στο Κοινοβούλιο, ως μέλος του Κοινοβουλίου και κατάφερα να μάθω κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Όταν θέλουμε εδώ να απευθύνουμε μία, μία ομιλία, θα πρέπει τουλάχιστον τρεις γλώσσες να χρησιμοποιούμε, γιατί δάλλως δεν βγαίνει. Γι' αυτό λοιπόν ε, σήμερα θα μιλήσω και γερμανικά και γαλλικά. Τα γαλλικά με δυσκολεύουν βέβαια, γιατί καταλαβαίνω τη γλώσσα, αλλά για να απευθύνω ομιλία στα γαλλικά ζορίζομαι. Θα συνεχίσω λοιπόν στα αγγλικά. Και γιατί είναι η τέταρτη γλώσσα μάλιστα. Μιλάμε για μια αλλαγή. Το τέλος της θητείας, οι υπερχόμενες εκλογές αποτελούν πραγματικά μια περίοδο περισυλλογή. Προτού όμω ε, κοιτάξουμε στο μέλλον, θέλω να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή για να το θέσουμε όλα αυτά στο σωστό πλαίσιο. Λετωνία, λοιπόν. Ευρώπη. Τι ενώνει τους Ευρωπαίους. Η κοινή ιστορία από την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Ρώμη, μέσω του χριστιανισμού που διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη και ο χριστιανισμός και ο πολιτισμός διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη και τελικά τα τελευταία προπήργια ήταν οι βαλτικές χώρες, οι οποίες ακόμα δεν είχαν προσαρτηθεί σε αυτόν τον κοινό χώρο, τον πολιτισμικό και θρησκευτικό, σε ό,τι αφορά την πολιτιστική και την θρησκευτική αυτή κληρονομιά. Μόλις στην 13ο αιώνα ο Παπάς είπε ναι σε μία σταυροφορία στις βαλτικές χώρες για τους μη χριστιανούς. Και έκτοτε η χώρα μας πέρασε όλες τις ε, πολιτισμικές εξελίξεις ε, και αναστατώσεις ε, που πέρασε και η υπόλοιπη Ευρώπη, τη μεταρρύθμιση, την αναγέννηση, το διαφωτισμό. Σήμερα η χώρα μας είναι λουθερανική κατά μεγαλύτερο βαθμό στο νότο και το ανατολικό κομμάτι πιο πολύ. Και θεωρούμε τον εαυτό μας μέσω της ιστορίας μας ήμασταν τμήμα του βορειοευρωπαϊκού πολιτισμικού χώρου και αυτό το λέμε με ρεαλιστικό τρόπο. Είμαστε ρεαλιστές, υπομονετικοί και θέλουμε να είμαστε πάντα μετριοπαθείς. Έχουμε μεγάλη δημιουργικότητα, μεγάλη επιχειρηματικότητα. Αυτό πάντα μας διεκρινέ. για εκατοντάδες χρόνια μετά την εισαγωγή και την... το χριστιανισμό στη χώρα μας. Αντιμετωπίσαμε διάφορες πολιτικές και στρατιωτικές αναστατώσεις από την Γερμανία, από την Πολωνία ενίοτε, από τη Σουηδία και άλλες φορές από τη Ρωσία. Σε όλη αυτή την φάση διατηρήσαμε την ταυτότητά μας και τη γλώσσα μας βέβαια. Και μόλις στα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 1918 διακηρύξαμε την ανεξαρτησία μας επιτέλους. Πήρε άλλα δύο χρόνια ο πόλεμος της ανεξαρτησίας ε, να απελευθερώσει την χώρα από τα στρατεύματα τα γερμανικά και τα ρωσικά που ήταν στην ε, χώρα μας. Και ο παππούς μου, σε ό,τι αφορά την προσωπική μου ιστορία, μπήκε στον τσαρικό στρατό ως στρατιώτης ε, του Τσάρου και έγινε μετά πολσεβίκο στρατιώτης κατά της του Τσάρου και όταν άκουσε ότι η χώρα μα ανακήρυξε την εξαρτησία τη, έγινε πολεμιστή τη ελευθερία, υπέρ τη ανεξαρτησία. Και αυτό αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα τη εποχή. Η χώρα μα αναπτύχθηκε λοιπόν μεταξύ των πολέμων στο Μεσοπόλεμο και μετά ήρθε και ο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεγάλε μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στην Ευρώπη και εδώ μπήκα και εγώ στην ε, εικόνα αυτή. Εγώ είμαι γιος μεταναστών του πολέμου το 1944 οι γονεί μου ήταν 18 και 14. Έφυγαν από τη Λετωνία στη Σουηδία. 5.000 περίπου Λετωνοί έφυγαν στη Σουηδία και κάποιοι πιο λίγοι στη Γερμανία όταν ο Σοβιετικός στρατός ερχόταν για δεύτερη φορά να καταστρέψει τη χώρα. Οι γονεί μου λοιπόν μεγάλωσαν στη Σουηδία, γνωρίστηκαν, παντρεύτηκαν και μετανάστευσαν στη ΣΥΠΑ όπου γεννήθηκα κι εγώ μαζί με τις δύο αδερφές μου. Πρώτα ήρθα μάλλον και πρώτη φορά στη Λετωνία το 1984. Τότε ήμουν ε, μαθητή στο Λύκειο, στο τελευταίο σχολείο μεταναστών ε, στη Γερμανία για Λετωνού. Τότε για πρώτη φορά πήγα στη Λετωνία και ο κόσμο τότε ήταν διαφορετικό. Η χώρα ήταν διαφορετική, η ώρα ήταν γκρίζα. Ο κόσμο δεν γελούσε, δεν χαμογελούσε στον δρόμο. Σοβιετικοί στρατιώτε παντού. Όλα στα ρωσικά υπήρχε πραγματικά έλλειψη επενδύσεων σε οποιαδήποτε υποδομή, κτίρια, δρόμους, ε, γέφυρες. Πραγματικά αποσύνθεση επικρατούσε. Και όταν ξεκίνησε η αλληλεγγύη στο τέλος του, της δεκαετίας του 80 και έπεσε και το τείχος του Μερολίνου στο 89, ξεκίνησε η αλλαγή. Το 91 επιτέλους ε, αποκτήσαμε την εξαρτησία μας και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αναπτύξαμε δημοκρατικούς θεσμούς. Αναπτύξαμε ελευθερή επιχειρηματικότητα, τραπεζικό σύστημα, οικονομία της αγοράς, από το τίποτα, από το μηδέν. Το 2004, 13 μόλις χρόνια μετά την ανεξαρτησία μας, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Μέσα σε λίγες εβδομάδες θα γιορτάσουμε τα 15 χρόνια από την προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ να σας πω εξ ονόματος της χώρας μου ολόκληρη ότι δεν έχουμε μετανιώσει την προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε μία ημέρα. So what, what is, what is the EU? Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πρώτα πρώτα, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, είναι μια ένωση αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου ιστορικά στην Ευρώπη. Πώς λύνονταν οι διαφορές. Με όπλα, με στρατιώτες, με τάγκς, με καταστροφή. Σήμερα πώς λύνουμε τις διαφορές. Με κουραστικές συζητήσεις, ε, διαφωνίες, ψηφοφορίες, αλλά με τρόπο διαφορετικό από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και σαν στόχο την οικονομική ανάπτυξη και στο κέντρο της είναι η ενιαία αγορά. Ανοίγοντας τα σύνορά μας, οι μεν στου δε, δημιουργήσαμε μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. 500 εκατομμύρια άτομα που πάνω κάτω είναι αντίστοιχη αγορά με αυτή τον ΙΠΑ που θεωρείται η ισχυρότερη οικονομία. Τα πράγματα ωστόσο δεν είναι όλα καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι γνωρίζουμε ως πολιτικοί ότι υπάρχει ισχυρό αντιευρωπαϊκό αίσθημα. Υπάρχουν πολιτικοί που παρέχουν απλουστευτικές απαντήσεις σε σύνθετα, πολύ σύνθετα ζητήματα. Τους χαρακτηρίζουμε γενικά ως λαϊκιστές. Με απλά μηνύματα, ε, το, το μήνυμά μου είναι μην ε, πολεμάτε τους λαϊκιστές, αλλά αντίθετα ακούστε γιατί ο κόσμος ακούει Προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί ο κόσμο ακούει του λαϊκιστέ και είναι δυσαρεστημένο. Πηγαίνετε λίγα χρόνια πίσω, 2008-2009. Μία τράπεζα κατέρευσε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Καταραίων που και που. Αυτό οδήγησε σε μια αλυσιδωτή αλλαγή τραπεζικών κρίσεων ανά τον κόσμο, ιδίω στην Ευρώπη, που οδήγησε σε μια οικονομική κρίση. Τη μεγαλύτερη μετά την κρίση του 1929 το ΑΕΠ της χώρας μου έπεσε σχεδόν κατά το 1 τέταρτο και σε άλλες χώρες μειώθηκε το ΑΕΠ ίσως όχι τόσο πολύ. Βγαίνοντας από την οικονομική κρίση, τι συνέβη λίγα χρόνια μετά, η μεταναστευτική κρίση, η ανασφάλεια, η, η, η πόλεμη στην Μέση Ανατολή οδήγησε σε μετακινήσεις πλησμών, πρόσφυγες και μετανάστες. Αποτέλεσμα είναι αυτό που εγώ χαρακτηρίζω ως πολιτική κρίση. Ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του στο σύστημα. Είναι κατανοητό αυτό. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να ξανααποκτήσουν την εμπιστοσύνη τους. Αν δείτε τους ε, ψηφοφόρους, θα δει ποιες είναι οι βασικές τους ανησυχίες. Τέσσερις θα έλεγα. Δουλειές, τρόπος ζωής, μετανάστευση, περιβάλλον και ασφάλεια. Για να μιλήσουμε για το μέλλον στην Ευρώπη πρέπει να μιλήσουμε για τα τέσσερα αυτά θέματα. Δουλειές πρώτα-πρώτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν μηχανισμό για ταχύτερη ανάπτυξη των θέσεων εργασίας. Αυτό που αποκαλούμε ενία αγορά. Θυμάμαι μια ιστορία όταν ήμουν παιδί. Μπορεί να είναι ένας μύθος του εσώπου, δεν ξέρω. Ένα παιδί, είχε, ε, ένας πατέρας είχε τρία παιδιά. Δίνει ένα μπαστούνι στον ένα και του λέει σπάστο. Και το παιδί το σπάει. Το δίνει στο δεύτερο και στον δεύτερο και του λέει σπάστο. Το σπάει και αυτό. Και στον τρίτο του δίνει ένα πακέτο με, μπαστού, με, με, με μπαστούνια και του λέει σπάστα και αυτός δεν μπορεί να τα σπάσει. Το, δι, το, το, αποτέλεσμα, το, το, το ηθικό δίδαγμα από αυτό είναι ότι όταν είσαι μόνος σου σπάς εύκολα, όταν είσαι ενωμένο, είσαι ισχυρός και αυτό είναι το θετικό της ενίας αγοράς. Έχουμε μια σειρά προκλήσεων για την ενία αγορά απ' έξω η άνοδος της Κίνας. Η, μια κυβέρνηση τον είπα, που δεν πιστεύει τόσο πολύ ότι μπορεί να παίξει πλέον ένα μείζωνα ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και στο παγκόσμιο εμπόριο. Κίνα πρώτα. Είναι μια χώρα που ανοιχτά επιδοτεί τις τεράστιες βιομηχανίες της, οι οποίες έρχονται στην Ευρώπη και ανταγωνίζονται χω, με συγκριτικό πλεονέκτημα. Τι απαντάμε εδώ. Η απάντηση στον αθέμητο ανταγωνισμό, λέω, δεν είναι ο προστατευτισμός. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο των Κινέζων. Δεν θα πρέπει να γίνουμε σαν τους Κινέζους, να ζητήσουμε από τους Κινέζους να γίνουν σαν και εμάς, ανοίγοντας την αγορά τους. Έχουμε πολύ ισχύ ως Ένωση και ως ενία αγορά. Αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Όχι σαν μικρά μπαστούνάκια, αλλά σαν ένα, ένας βεσμός από ε, κράτη που μπορούν να επηρεάσουν τον κόσμο. Τώρα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάποια εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε, που σχετίζονται με τα εσωτερικά εμπόδια στην ενιαία αγορά. Ιδίως στην ψηφιακή σφαίρα και στις υπηρεσίες αναρωτηθείτε όπως αναρωτιέμαι και εγώ. Γιατί οι μεγαλύτερες εταιρείες του ίντερνετ προέρχονται από τις Ηνωμένε Πολιτείε και δεν είναι ευρωπαϊκές. Η απάντηση είναι προφανής. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχει μια ζώνη δολαρίου, μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ομοσπονδιακό προπολογισμό και μηδενικά εμπόδια μεταξύ των πολιτιών στο εμπόδιο. Έχουν μια πραγματικά ενωμένη ενιαία αγορά, μικρότερη από εμά, 330 εκατομμύρια κατοίκου. Έχουμε μεγαλύτερη αλλά πολλά εμπόδια. Όταν λοιπόν λέμε ότι θέλουμε να έχουμε εθνικούς πρωταθλητές, δεν θα πρέπει να κάμπτουμε την ε, νομοθεσία για τον ανταγωνισμό για να δημιουργούμε τεχνητά εθνικούς ε, πρωταθλητές, αλλά να μειώνουμε τα εμπόδια στο εσωτερικό της αγοράς για να αναπτυχθούν πραγματικά αυτοί οι πρωταθλητές και να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ένας από τους ακρογωνιαίους λήθους της ενίας αγοράς είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τράπεζες. Πριν από 10 χρόνια η μεγαλύτερη απειλή εναντίον αυτών ήταν η ρευστότητα. Οπότε δημιουργήσαμε την Τραπεζική Ένωση έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Εντοκή Τράπεζα να επιτηρεί ε, τις πιο μεγάλες από αυτές. Από τότε όμως ο κόσμος έχει αλλάξει. Η ρευστότητα δεν είναι πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ένα νέο πρόβλημα προέκυψε που είναι η τρομοκρατία και η χρηματοδότηση τρομοκρατία στην Ευρώπη. Και πώ συμβαίνει αυτό πολύ συχνά μέσω παράνομων μεταφορών μέσω του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Οπότε πού είναι η νομοθεσία μας για το ξέπλυμα χρήματο. Με την κυρία Σαρτζεντίνη ήμουνα συνεισηγητής παλιότερα για αυτό το θέμα και έμαθα αρκετά πράγματα. Η νομοθεσία κατά του ξεπλήματος ε, χρήματος έχει σχέση, ε, άμεση σχέση με την αξιολόγηση κινδύνου και με την αποφυγή του βρώμικου, χρήματος να μπαίνει, ε, να, βρώμικο χρήμα να μπαίνει στο τραπεζικό μας σύστημα. Για τα τελευταία 20 χρόνια ποσά από την Ρωσία προσπαθούν να βγουν από τη Ρωσία. Γιατί, Γιατί η Ευρώπη είναι ασφαλής, έχει ασφάλεια δικαίου, κράτος δικαίου και κανείς δεν σου αρπάζει τα χρήματα ε, πολλά από αυτά τα χρήματα που έρχονται από τη Ρωσία είναι καθαρά, αλλά κάποια όχι. Αυτοί οι εγκληματίε που προσπαθούν να φέρουν χρήματα από τη Ρωσία στην Ευρώπη, δεν μιλώ για αυτού που προσπαθούν να ε, βελτιστοποιήσουν ε, το φόρο πληρών κλπ. Μιλώ για ανθρώπου οι οποίοι ε, θέλουν να φέρουν βρώμικο χρήμα. Αυτοί, σαν γεράκια, υπερίπτανται και προσπαθούν να βρουν του αδύναμου κρίκου στην αλυσίδα. Εδώ σε αυτή τη χώρα μπορεί να κάνει αυτό, σε εκείνη τη χώρα μπορεί να, δεις κάτι άλλο, να κάνει κάτι άλλο κλπ. Ε, και εμεί ήμασταν τμήμα αυτή τη αλυσίδα. Ε, το, όμως δεν είμαστε μόνοι μα. ε, το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Από τότε που έγινα πρωθυπουργό, δεν μπορώ να περιμένω όλοι να συμφωνήσουμε, οπότε εγώ καθαρίζω το σπίτι μου. Θα έχουμε το πιο καθαρό και ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη. Σε 1,5 χρόνο θα μπορούμε να σα ενημερώσουμε τον καθένα σα ε, ξεχωριστά και όλοι μαζί για το πώ μπορεί να καθαρίσει κανεί το τραπεζικό σύστημα. Θα διώξω τα ποντίκια από το δικό μου σπίτι. Και το δικό μου σπίτι θα είναι καθαρό. Αλλά τι θα γίνει με του γείτονε. Οι εγκληματίε μπορεί να εγκατέλειψαν τη Λετωνία, αλλά είμαι σίγουρο πω δεν εγκατέλειψαν την Ευρώπη. Οπότε θα πρέπει να ε, καθαρίσουμε όλη τη γειτονιά. Αυτό σημαίνει ότι η τραπεζική εποπτεία για την καταπολέμηση του, ε, του, του ξεπλήματος θα πρέπει να είναι βασική μας μέρημνα. Μια άλλη, μου, ε, μια άλλη ανησυχία των ψηφοφόρων είναι ο τρόπος ζωής του και η μετανάστευση. Εδώ δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις, δεν έχω εγώ απλές απαντήσεις και δεν νομίζω ότι κανείς έχει. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είναι ένας εξαιρετικό προορισμό για να ζει κανεί και να εργαστεί. Σταθερέ οικονομίε, σταθερέ δημοκρατίε κράτος δικαίου, ε, ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες, ενώ πολλοί από τους γειτονέ μας δεν έχουν κάτι τέτοιο. Οπότε οι πίεση, οι πιέσεις, ε, μεταστευτικές πιέσεις αυξάνονται. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα εξαλειφθεί, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Η χώρα μου δέχτηκε κάποια μετανάστευση. Πάνω από 700.000 άτομα μετανάστευση έφτασαν στη χώρα μου κατά τη διάρκεια του Σοβιετικού καθεστώτος. Το 1 τρίτο του πληθυσμού μα. Έτσι είμαστε 2 εκατομμύρια. Δεν είχαμε κυβέρνηση τότε, οπότε <laughs> δεν πήραμε εμεί αυτέ τι αποφάσει. Τι αποφάσει λαμβανόντουσαν από τη Μόσχα. Δεν υπήρχε διαδικασία συναπόφαση, δεν είχαμε λόγο. Με, αφού ανεξαρτοποιήθηκαμε, πώ το αντιμετωπίσαμε μέσω της ένταξης. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Πρέπει να συνεργαστούμε με αυτούς, να προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα έτσι ώστε αυτοί οι μετανάστες να ενταχθούν στη δική μας κουλτούρα. Αυτό είναι ο, ο μόνος τρόπος. Ε, δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει αυτό. δεν μπορεί κανείς να αποφύγει ότι κάποιοι θα θέλουν να έρχονται συνεχώς στην Ευρώπη. Θα πρέπει να τους εντάσσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να μετριάσουμε τις ροές είναι τα εξωτερικά σύνορα, η Frontex. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που πρέπει να ενισχυθεί. Αν αποδείξουμε στους ψηφοφόρους μας ότι ελέγχουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, μπορούμε να έχουμε ελεύθερα εσωτερικά σύνορα. Θυμάστε πόσο εύκολο ήταν παλιότερα ε, να κυκλοφορεί κανείς στη ζώνη του Σέγγεν ε, μεταξύ για παράδειγμα Στρασβούργου και Γερμανίας. Τώρα πια πολλές φορές οι γέφυρες κλείνουν, ξανά τοποθετούνται τα σύνορα. Ε, αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε ισχυρά εξωτερικά σύνορα και χρειαζόμα, χρειάζεται να χρηματοδοτήσουμε ε, ε, καταβλισμούς προσφύγων και μεταναστών. Χρειάζεται να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες και να τις χρηματοδοτήσουμε και οπωσδήποτε θα πρέπει να εργαστούμε πάνω στην ένταξη των μεταναστών. Είμαστε μια ένωση 28 ακόμα κυρίαρχων κρατών, το καθένα με τη δική του εθνική ταυτότητα, οπότε είναι εξαιρετικό, εξαιρετικά σημαντικό να διατηρήσουμε την κουλτούρα μας, τη γλώσσα μας και την εθνική μας ταυτότητα. Αυτό μέσω της ένταξης, της ενσωμάτωσης όσων έρχονται στη χώρα μας, στις χώρες μας και θα πρέπει να προσαρμοστούν. Σε αυτό θα πρέπει να εργαστούμε. Αν αποδείξουμε ότι ελέγχουμε τα εξωτερικά σύνορα και μπορούμε να εντάξουμε τους μετανάστες, οι ψηφοφόροι θα χαλαρώσουν σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Τρίτη ανησυχία τους, το περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή είναι αληθινή. Είναι κάτι το αληθινό ένα γεγονός ο άνθρακας και η ε, ορυκτή υδρογονάνθρακες εξακολουθούν να καίγονται και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Οπωσδήποτε θα πρέπει να πάρουμε πολλά μέτρα και επιλαμβάνουμε ε, ενεργειακή αποδοτικότητα κλπ. Το σημαντικό όμως είναι το ενεργειακό μείγμα. Εμείς είμαστε δεύτεροι μετά τη Σουηδία σε ό,τι αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, 45% του συνολικού μα μείγματο. Δεν είναι όλε οι χώρε έτσι. Πολλέ χώρε εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τον άνθρακα. Δεν μπορούμε όμω να μειώσουμε τη χρήση του άνθρακα με επιθυμίε, κάποιο πρέπει να πληρώσει αυτή τη μετάβαση και θα χρειαστεί χρόνο. Ανεξαρτητός όμως του πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε, υπάρχει μία διαστατική αλλαγή που πρέπει να γίνει έτσι ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση. Και πάλι αυτό είναι το άνοιγμα της ε, αγοράς ενέργειας στον ανταγωνισμό. Χρειάζεται ανταγωνισμός σε ανανεώσιμες. Για παράδειγμα, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλές χώρες ε, έχουν ρυθμίσει ε, το θέμα της ενέργειας, τον αγορά ενέργειας, οπότε οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο ανεξάρτητα από την ώρα τη ε, μέρα ή από τη μέρα τη εβδομάδα. Οπότε δεν σε νοιάζει. Μπορεί να βάλει το πλυντήριό σου να δουλέψει όποια στιγμή τη μέρα, όποια μέρα τη εβδομάδα θέλει. Όταν όμω ανοίγουμε τι αγορέ μα στον ανταγωνισμό, ή ο ανταγωνισμό ε, δίνει κίνητρα και αντικίνητρα με μειώσει τιμών ή αυξήσει τιμών ανάλογα με την ώρα τη μέρα, τη μέρα τη εβδομάδα. Οπότε μειώνουμε ε, τις ε, ανάγκες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες εχμής αν μπορούμε σε αυτές τις ώρες αιχμής, για παράδειγμα, να επιτρέψουμε στα ψυγεία να αυξήσουν θερμοκρασία τους κατά ένα-δύο βαθμούς, αυτό μας εξοικονομεί πάρα πολύ ενέργεια. Για αυτά τα πράγματα χρειαζόμαστε ανταγωνισμό και χρειαζόμαστε απορρίθμιση. Τέταρτη ανησυχία των πολιτών μας, η ασφάλεια. Αυτό σημαίνει κάτι διαφορετικό ε, για τον Νότο, διαφορετικό για τον Βορρά. Στο Νότο, όταν μιλάμε για ασφάλεια, ε, ε, το μυαλό πηγαίνει πιο πολύ στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση και στην τρομοκρατία. Στη Δυτική Ευρώπη, η μεγαλύτερη απειλή εναντίον της ασφάλειας είναι το ανεξέλεγκτο Brexit ενδεχομένως και για το εμπόριο αλλά και για την ειρήνη στην Βόρεια Ιρλανδία. Εγώ προέρχομαι από τη Λετωνία. Όταν εμείς έχουμε στο μυαλό μας την ε, μιλάμε για ασφάλεια, έχουμε στο μυαλό μας τη Ρωσία. Ε, αυτό είναι κοινό μυστικό. Ε, η Ρωσία είναι ένας γείτονας που έχει μια κυβέρνηση που έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Πιστεύει ότι περικυκλώνεται από εχθρούς που είναι έτοιμοι να τις επιτεθούν. Αυτό είναι το <laughs> αμυντικό δόγμα της Ρωσίας. Ε, οπότε προσπαθεί να αποδυναμώσει τους γειτονές της. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη απειλή από τη Ρωσία δεν είναι στρατιωτική. Και το στρατιωτικό είναι απειλή, αλλά δεν είναι η μεγαλύτερη απειλή. Έχουμε το ΝΑΤΟ, έχουμε τη δική μας προετοιμασία. Η μεγαλύτερη απειλή είναι τα ψεύδη και οι ψεύτικες πληροφορίε ή ψευδείς πληροφορίες, fake news. Ζούμε στον κόσμο αυτών των πολυόμορφων συσκευών, όλοι έχουμε από μία τουλάχιστον, Πίστευα, όπως όλοι μας παλιότερα, ότι θα μας ε, εξασφαλίσουν αυτές τις συσκευές απόλυτα ελεύθερη ε, πρόσβαση στις πληροφορίες. <laughs> Και γίνεται αυτό. Απ' την άλλη μεριά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένας τρομακτικά καλός τρόπος για την διάδοση ε, χωρίς καμία καθυστέρηση ε, ψευδών ειδήσεων. Και όλο και περισσότερος κόσμος εγκαταλείπει ε, τη, αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους υπεύθυνους δημοσιογράφους που ελέγχουν τις πληροφορίες κλπ. και πιστεύει, ε, πέφτει θύμα ψευδών πληροφοριών που διαδίδονται μέσα στο διαδίκτυο. Οπότε έχουμε ευθύνη για τις πλατφόρμες που ε, διαδίδουν στο ίντερνετ αυτές τις πληροφορίες. Προφανώς είναι ολιστηρός ο δρόμος, γιατί είναι πολύ λεπτή η γραμμή ανάμεσα στην ε, ευθύνη ε, και ε, στη φήμωση, στη λογοκρισία. Δεν θα υποστηρίξω ποτέ τη λογοκρισία, αλλά θα πρέπει να βρούμε το όριο. Γιατί πρέπει να δούμε τι προσπαθούν να κάνουν. Προσπαθούν να διχάσουν την κοινωνία, να μας ε, φέρουν σε σύγκρουση μεταξύ μας. Για παράδειγμα, εμβολιασμοί. Από πού ξεκίνησε το επιχείρημα ότι οι εμβολιασμοί οδηγούν σε αυτισμό. Οι Ρώσοι ξεκίνησαν αυτή, αυτό τον ισχυρισμό. Και η, ε, η αποφυγή του εμβολιασμού δημιουργεί πολλά προβλήματα στην Ευρώπη. Μετανάστευση και στη μετανάστευση πολλά τα ψεύδι που ξεκινούν από τη Ρωσία, το Brexit. Έχει γίνει, ο Τζορτ Σόρος έχει γίνει μια φούσκα στην Ανατολική Ευρώπη ότι δήθεν ε, συνωμοτικά επηρεάζει τη ζωή όλων μας κλπ. Αν δεν δεχτούμε το, την πραγματικότητα δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Η, για την ασφάλεια ε, η στρατιωτική απειλή δεν είναι τόσο μεγάλη. Ε, Παρ' όλα αυτά, εμείς επενδύουμε 2% του προπολογισμού μας στην ασφάλεια και, όλοι, όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να κάνουν το ίδιο. Απ' την άλλη μεριά, εξίσου σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ψευδών ειδήσεων. Και εκεί μάλλον θα πρέπει να εξετάσουμε το κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει μέσω νομοθεσία. Τέλος, ε, έχω και κάποια θέματα σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέλω να, ε, τα οποία θέλω να σας σχολιάσω. Πρόκειται για τον 7ετή προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνο, όπως και εσείς, ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην έρευνα και τεχνολογία στην Ευρώπη. Έχουμε πολλούς νέους έξυπνους ευφύς ανθρώπους που θα πρέπει να τους κρατήσουμε στην Ευρώπη και να τους αναπτύξουμε εδώ. Όμως, εξίσου σημαντικό είναι αυτή η επένδυση να μην γίνεται μόνο σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Γιατί έξυπνα με μυαλά υπάρχουν παντού στην Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη χρειάζεται επένδυση στην αριστεία. Η αριστεία δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο σε 2, 3, 4, 5 πρωτεύουσε. Ναι, λοιπόν, στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να διαχυθεί σε όλη την Ευρώπη. Η ευφυή συνοχή. Η συνοχή εξακολουθεί να είναι ε, σημαντική, αλλά θα πρέπει να είναι ευφυή. Θα πρέπει οι πιο φτωχέ περιοχέ να συγκλίνουν προ τι πιο πλούσιε. Αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε. Τέλο, το θέμα των αγροτών στην Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό παλιότερα αφιερωνόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ΚΑΠ. Όχι τόσο όσο παλιά, αλλά εξακολουθεί αυτό το φαινόμενο και σήμερα. Είναι ιστορική ευκαιρία μας να ε, εξαλείψουμε μια ιστορική αδικία. Αυτή τη στιγμή επιδοτούμε μέσω άμεσων πληρωμών τους γεωργούς μας. Υπάρχει όμως μια παγίδα. Οι επιδοτήσεις δεν είναι ισότιμες, παρόλο που τα προϊόντα τους διατίθενται με ισότιμους τρόπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που είναι λιγότερο ευνοημένοι είναι οι βαλτικές χώρες. Για μαθηματικούς λόγους που σχετίζονται με τα δεκαετία του 90, εμείς επιδοτούμαστε λιγότερο σε σχέση με άλλους. Οι δικοί μας γεωργοί ανταγωνίζονται με ίσους όρους με τους υπόλοιπους γεωργούς, αλλά αυτό θα ήταν πραγματικά ισότιμο αν επιδοτούνται με τον ίδιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να μειώσουν, να χαμηλώσουν το βιωτικό τους επίπεδο για να μπορούν να ανταγωνίζονται με θεμητό τρόπο. Αν συνεχίσουμε την επιδότηση, η επιδότηση αυτή θα πρέπει να είναι ισότιμη για όλους. Τελειώνω, μπορείτε να αναπνεύσετε. Τάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άριστη, δεν είναι τέλεια, ούτε και θα είναι στο μέλλον. Αλλά είναι το καλύτερο πόσα θα μπορούσα να φανταστώ. Στην Ευρώπη, για εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα χρόνια, οι διαφορές ρυθμιζόντουσαν ε, με την δύναμη του πιο ισχυρού. Ποιος είναι ο πιο ισχυρός, αυτός επικρατεί, ο πιο αδύναμος, κρίμας, πρόσεχε. Τώρα πια εργαζόμαστε με διαφορετικό τρόπο, με έναν τρόπο που είναι καλύτερο από οποιονδήποτε άλλο είχαμε φανταστεί ποτέ στην ιστορία μας. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε και αποφασίζουμε ε, με δική μας βούληση και με την επιθυμία των πολιτών μας. Κάποιο μπορεί να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το Brexit αποδεικνύει πόσο δύσκολο είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, αποτελεί μαρτυρία του πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καλή θέληση και η, συνένεση να παραμείνουμε σε μια Ευρώπη των 27 αποτελεί μαρτυρία και απόδειξη ότι είμαστε πεπισμένοι πως μέσω συζήτησης, μέσω του διαλόγου μπορούμε να παραμείνουμε ενωμένοι και να προχωρήσουμε χωρίς ε, να χρησιμοποιούμε βία, χωρίς να προσφεύγουμε στη βία. Μιλώντας ο με τον άλλο. Τώρα για το μέλλον. Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα βασικά. Την ενία αγορά. Να καταργήσουμε τα, τους φραγμούς. Να ελέγξουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα. Να μειώσουμε τον, την απειλή της ανεξέλεγκτης ε, μετανάστευσης. Ε, ευφύης μετάβαση στις, ε, ε, μορφές ενέργειας. Ε, ενίσχυση της ασφαλείας μας, όχι μόνο στο στρατιωτικό σκέλος, αλλά και στην ασφάλεια της πληροφορίας. Μην πολεμάτε τους λαϊκιστές. Αντιμετωπίστε την ουσία και τον λόγο της αιτίας της ανησυχίας των πολιτών. Θυμηθείτε το μύθο αυτό του Εσώπου ε, με τις βέργες που είναι δύσκολο να τις πάσει κανείς όταν είναι μια θυμονιά. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ισχυρό παίκτη ε, στον κόσμο και έχουμε βασικέ αξίε. ελευθερία, δημοκρατία, κράτο δικαίου και αυτέ θα πρέπει να προβάλλουμε και στι άλλε χώρε του κόσμου. Ευχαριστώ. Ε, είστε πολύ δημοφιλής, ε, αγαπητέ κύριε Κριστιανής. Αγαπητέ Κριστιανής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν και έχει το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Χαίρομαι που ξαναβλέπω εδώ τον Πρωθυπουργό της Λετωνίας, που γνωρίζει πολύ καλά το ημικύκλιο γιατί ήταν ευρωβουλευτή για εννέα έτη. Τον χαίρο, χαίρο ιδιαίτερα που τον βλέπω γιατί θυμάμαι πάντα την λετονική προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών και θυμάμαι την προεδρία γιατί ήταν η πρώτη πραγματική προεδρία επί επιτροπής μας. Συνυπάρξαμε για δύο μήνες με την Ιταλική Προεδρία. Θυμάμαι την τελευταία μέρα της προεδρίας αυτής της Λετωνίας. 29 προς 30 Ιουνίου νύχτα υιοθετήθηκε η οδηγία για τα roaming, για τα τέλη περιαγωγής, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην τηλεφωνία και το ίντερνετ. Κάτι που αποδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί να πετύχει και πρέπει να κρατάμε την ελπίδα μας μέχρι τελευταία μέρα συχνά συζητούμε, σαν να μην είχαμε άλλο πράγμα να κάνουμε για το Brexit. Πριν τι εκλογέ θα ήταν, θα ήταν ίσως σκόπιμο να τονίσουμε προ τους πολίτες τι επιδόσεις της Ένωσης τα τελευταία χρόνια. ιδίω την χρήσιμη απόφαση για την περιαγωγή. Σημαντικό είναι το Brexit, σημαντικότερη η καθημερινότητα των πολιτών. θελήσαμε να είμαστε και γίναμε η Επιτροπή του Διαλόγου. Οργανώσαμε συναντήσεις με τους πολίτες. 1.600 συναντήσεις διαλόγου με τους πολίτες. Κάτι που αποδεικνύει ότι οι επίτροποι δεν κλείνονται στα μπούνκερ του και κυκλοφορούν ανά την Ευρώπη. Αυτό αποδεικνύει ότι η Επιτροπή δεν είναι μια συμμορία πραξικοβηματιών χωρίς νομιμοποίηση, αλλά είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει χωρίς να το θέλουν οι πολίτες, χωρίς τα έθνη. Τα έθνη είναι σημαντικά. Αυτοί που πιστεύουν ότι τα έθνη είναι μια προσωρινή δημιουργία της ιστορίας, σφάλουν. Οι, τα έθνη έχουν διάρκεια δεν πρέπει λοιπόν να μιλάμε για Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη πλέον, διότι δίνει την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται κράτο ή Η Ευρώπη δεν θα γίνει ποτέ ένα κράτος που θα αντιγράψει το μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτείων τη Ευρώπη. Είστε Λετωνός, Βαβαρός, Βρετόνος, Γάλλος, Λουξεμβουριέζος και Ευρωπαίος. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στον πατριωτισμό αν ο πατριωτισμός είναι υπεύθυνο και αντιλαμβάνεσαι την ανάγκη, την συμμετοχή σε ένα ευρύτερο σύνολο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ως Επιτροπή θελήσαμε να πάψουμε να παρεμβαίνουμε σε όλα τα μικρά γεγονότα της καθημερινότητας των πολιτών και να στραφούμε στα μεγάλα ζητήματα που διακυβεύονταν στο μέλλον. Αυτό ήταν και η συμφωνία που είχαμε κάνει μαζί σας, τους εκπροσώπους των λαών της Ευρώπης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχα υποβάλει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της Επιτροπής μας. Δεν ήταν ε, λόγια του αέρα. Είχαμε υποβάλει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που προωθήσαμε ήδη την πρώτη χρονιά. Μέχρι σήμερα. 350 από τις προτάσεις μας έχουν εγκριθεί ενώ 164 παραμένουν ακόμα στην τράπεζα του, στο τραπέζι των συνομοθετών. Εγώ θα είχα βέβαια ε, την επιθυμία να προχωρήσουν όλες οι μεταρρυθμίσεις που είχαμε προτείνει για το καθεστώς του ασύλου, για παράδειγμα. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι ποτέ δεν είχαμε τόση πολύ πρόοδο στα κοινωνικά ζητήματα που για πολλά χρόνια ήταν ο φτωχός συγγενής της ανάπτυξης της Ευρώπης. Αυτό θα έπρεπε να... Αυτό άλλαξε και, προ... και τώρα η, προσπάθεια του, της Επιτροπής είναι ακριβώς να συνοδεύονται οι δύο κατηγορίες. Η Λετωνία είναι μια χώρα που αξίζει και άξιζε την συμμετοχή της στην Ένωση, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργό της Λετωνίας πριν από λίγο λόγια. Είχα, είπατε, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι όντως η χώρα σας ανέλαβε τις ευθύνες της και πραγματικά όπως λένε οι ποιητές σας, ε, θα, θα, θα είμαστε τόσο μεγάλοι όσο μπορούμε, όσοι θέλουμε να είμαστε. Και αυτό το πετύχατε. Αγωνιστήκατε για την ελευθερία σας κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από αυτές που φαντάζονταν οι Δυτικοευρωπαίοι. Κάνατε ιστορία αντί να υποστείτε πίεση από τους μεγάλους, όταν υποστήκατε τις πιέσεις από τους μεγάλους γείτονές σας. Είπατε όχι στα όπλα. Επιδιώξατε με ειρηνικό τρόπο την ελευθερία σας. Και αποτελείτε, και αυτό αποτελεί ένα από τα καλύτερα συμβάντα της σύγχρονης ιστορίας. Ο τρόπο με το οποίο η Λετωνία και οι άλλες βαλτικές χώρες αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία τους. Η Λετωνία δεν έχει θέση στο σκοτάδι, στη σκιά, αλλά στον ήλιο, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά μια μεγάλη μέρα η μέρα στην οποία η Λετωνία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπήκαμε στην, ε, μπήκατε στην, ε, στο Σέγγεν και σύμφωνο απόλυτα με αυτά που είπατε για τα ιστορικά σύνορα και την, ε, τα ιστορικά σύνορα. Την ασφάλεια αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ακτοφυλακή, συνοριοφυλακή με 10.000 ε, προσωπικό, άντρες και γυναίκες. Το Συμβούλιο ήθελε να αναβάλει την πρόταση αυτή για το 2027. Ζητήσαμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020. Όλοι όμως λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Ας το κάνουμε λοιπόν πραγματικότητα. βοηθάτε να καταστεί η Ευρώπη πιο δυνατή και πιο ασφαλής. Είσαστε ένα από τα 25 κράτη-μέλη που ξεκίνησε την συνεργασία στα θέματα άμυνας τον Δεκέμβριο του 2017 και χαίρομαι που διαδραματίζεται σημαντικό ρόλο και σε άλλα σημαντικά θέματα σε ό,τι αφορά την στρατιωτική κινητικότητα και τη διευκόλυνση αυτής. Είναι σημαντικό αυτό για τη Λετωνία, η στρατιωτική κινητικότητα καθιστάτε λοιπόν ε, την κινητικότητα αυτή πιο εύκολη και κοιτάξτε, κοιτάξτε και το θέμα των ε, ζητημάτων αυτών και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει και ενισχύει την ενεργειακή επικυριαρχία και την εθνική επικυριαρχία. Κοιτάξτε τα θέματα ενέργειας, για παράδειγμα, που αποτελούν σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής, την ιστορία σας και τη γεωγραφία σας, που σημαίνουν ότι η Λετωνία και η Βαλτική ήταν αποκομμένοι από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αναλάβαμε τα καθήκοντά μας λοιπόν και τότε ξεκαθαρίσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αφήσει σε καμία περίπτωση τους πολίτες της να κρυώνουν και στο σκοτάδι. Για μένα αυτό τότε ήταν θέμα της Βαλτικής, ναι, αλλά όχι μόνο θέμα της Βαλτικής, αλλά ήταν και ευρωπαϊκό ζήτημα. Και γι' αυτό λοιπόν όταν αλάβαμε τα καθήκοντά μας ιδρύσαμε μια ενεργειακή ένωση και τη βάλαμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας για να μπορέσει και η Βαλτική και η Λετωνία και οι υπόλοιπε Βαλτικές χώρες να δουν ότι οι ενεργειακέ του ανάγκε καλύπτονται. Σήμερα λοιπόν εξυγχρονίζουμε την αγορά του ηλεκτρισμού. Μέχρι το 2025 επενδύουμε σε υποδομές και έχουμε την πιο φιλόδοξη πολιτική σε όλο τον κόσμο σε ό,τι αφορά την ενέργεια και το κλίμα. Είμαι ευτυχής που αυτή η αυτό το όραμα της Ενεργειακής Ένωσης υλοποιήθηκε και κατέστη πραγματικότητα και ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την ηγεσία του και για τη δουλειά που έκανε ως Πρωθυπουργό σήμερα και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο παρελθόν. Κύριε Πρόεδρε, αλλάζω γλώσσα. Η Λετωνία συμβάλλει στην Ευρώπη. Αυτό θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι φυσιολογικό και η Ευρώπη να επενδύσει στην Λετωνία γιατί επένδυση στη Λετωνία είναι επένδυση στο ευρωπαϊκό μέλλον. Οι Λετωνοί γνωρίζουν από πρώτη χέρι τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό. 50.000 ε, Λετωνοί αναζητούν δουλειά από το 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητούν επίση νέε δεξιότητε, νέε ικανότητε για να μπορέσουν να απορροφηθούν από την αγορά εργασία. 300 χιλιόμετρα νέα κτίρια και νέοι δρόμοι χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους για να συνδέσουν και, τις, ε, και να αναπτύξουν και τις ε, αστικές περιοχές αλλά και την Ήπεθρο στη Λετωνία. 960 δισεκατομμύρια επενδύσεις στη Λετωνία κινητοποιήθηκαν. Το μέλλον της Λετωνίας λοιπόν αφορά όλους μας, είναι το μέλλον όλων μας και γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε στον επόμενο προϋπολογισμό 100 δισεκατομμύρια ευρώ στην καινοτομία και στην έρευνα να επενδυθούν. Θέλουμε να επενδύσουμε στο μέλλον της Ευρώπης γιατί μόνο από κοινού και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Για παράδειγμα, θα τριπλασιαστούν ε, οι επενδύσεις στην ασφάλεια και θέλουμε επίσης και στο θέμα να υποστηρίξουμε τα, τους πόρους και τις επενδύσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, το Erasmus Plus. Διπλασιάζονται οι πόροι μάλιστα για το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του για την διαρκή υποστήριξη και την ενεργή συμμετοχή του. Να κάνω κάποιες ε, Παρατηρήσει όμω και σε ό,τι αφορά τι μεσοπρόθεσμε επενδύσεις και τον προγραμματισμό. Όντως, στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στην νεολαία επενδύουμε. Όλα αυτά όμως μπορούμε να τα κάνουμε μόνο αν γίνουν περικοπέ σε άλλες πολιτικές, συνοχή και σε γεωργία. Αυτό δεν με ικανοποιεί σε καμία περίπτωση, αλλά αν αφήσουμε τα πράγματα όπως έχουμε και προσθέσουμε και τι νέε προτεραιότητες, καπάκι, επί των οποίων συμφωνήσαμε, πολύ απλά θα καταρρεύσει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στο επίπεδο του 1,4%. Αυτό δεν το θέλει κανεί. Εμένα δεν θα με ενοχλούσε καθόλου, ξέρετε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αξίζει παραπάνω από 1,4% του ΑΕΠ της. Αλλά ακόμα και το ίδιο το Κοινοβούλιο σε θέματα δημοσιονομικά είναι λιγότερο διστακτικό μεν από το Συμβούλιο, αλλά ω ανώτατο όριο για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό έφτασε το 1,3%. Αν εμείς ε, από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνουμε 1,4%. Ούτε ακόμα και εσείς στο Κοινοβούλιο δεν θα συμφωνούσατε με το 1,4%. η γεωργία και η συνοχή είναι πολύ σημαντική τομεί και για κάποιες χώρες πιο σημαντική από ό,τι για άλλες βέβαια. Η Λετωνία έχει σημαντικά χρόνια, σημαντικό παρελθόν, όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής ε, της θέσης, αλλά και της ε, ιστορίας της, αλλά και λόγω των οικονομικών κρίσεων που έπληξαν την Λετωνία. Πέντε χρόνια ωστόσο μετά την ε, έναρξη της αντιμετώπισης της κρίσης η Λετωνία τα πηγαίνει καλύτερα. Και αυτό αποτελεί και επίτευγμα του προκάτοχου σας, του κυρίου Βαλτίς Ντομπρόφσκι, του προκατόχου σας, ο οποίος έθεσε στη σωστή πορεία τη Λετωνία. Και γι' αυτό κατέβαλα ιδιαίτερες προσπάθειες ε, να καταστεί εκ νέου επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για θέματα νομισματικά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλντής. Πολλά λοιπόν θα είχα να πω για αυτά που μας παρουσίασες. Μίλησες πάρα πολύ ώρα όμως και έτσι αναγκαστικά εγώ θα πρέπει να κλείσω σιγά σιγά. Η Λετωνία είναι μικρή χώρα και εγώ είμαι ειδικό στις μικρές χώρες, ξέρετε. Είναι όμως μια χώρα με μεγάλες φιλοδοξίες. Είναι το μέρος όπου συναντιέται η Ανατολή με τη Δύση. Δεν μπορεί η Ανατολή και η Δύση να διχάζονται. Είναι οι δύο πνεύμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν η Ευρώπη θέλει να έχει ένα καλό ε, μέλλον, θα πρέπει να αναπνέει και με τους δύο πνεύμονες της. Είναι η τελευταία αυτή ομιλία που απευθύνω προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βαριά καρδιά. Βλέπω ότι μερικοί συνάδελφοι αποχωρούν από την πολιτική και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά εδώ στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έμαθα πολλά, τσακώθηκα πολύ, αλλά θεωρώ ότι πετύχαμε και πολλά. Είχα πει την πρώτη μέρα της ε, των καθηκόντων μου η Ευρώπη είναι κάτι το οποίο πρέπει να ζήσει κανείς. Αν δεν τη ζήσουμε, δεν ζει η αγάπη μας ε, αυτή για την Ευρώπη. Εγώ αγαπώ την Ευρώπη και ε, μακάρι να ζήσει καλά η Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της ε, Κομισιόν, αγαπητέ Ζων Κλοντ. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία μας, παρόλο ότι μερικές φορές είχαμε και κάποιες πιο... Ε, είχαμε μερικές στιγμές έντασης στις συζητήσεις μεταξύ της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Για τα πιο σημαντικά όμως θέματα ε, εργαστήκαμε μαζί προς όφελος και προς συμφέρον των πολιτών μας, των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε ανάγκη την Ευρώπη. Προφανώς χρειάζεται να τη βελτιώσουμε, να την αλλάξουμε. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος ε, έτσι ώστε η Ευρώπη να προστατεύσει, να περαμηθεί της Ευρώπης και να προστατεύσει τους πολίτες της. Θυμάστε τι έγινε πριν από μερικέ μέρες στην Παναγία των Παρισίων. Ε, η, η γενικευμένη θλίψη που προέκυψε απέδειξε ότι έχουμε μια κοινή ψυχή, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες παρόλο που μπορεί να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για το έργο σου, για την προσήλωσή σου, για το πάθος σου και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε στο Συμβούλιο βέβαια. Ε, αλλά χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα και όλες τις προηγούμενες φορές. Συγχαρητήρια. Πρέπει να κλείσουμε ε, την εγγραφή για το Catch the Eye. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βέμπερ. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ σπουδαία ομιλία και να ευχαριστήσω τον ε, Πρόεδρό μας που διοργάνωσε αυτή την ομιλία στα πλαίσια του μέλλοντο τη Ευρώπη και χαιρόμαστε που Κριστιανή είσαι εδώ μαζί μα ω τελευταίο ομιλητή εδώ στην Ολομέλεια. Πολύ μεγάλη η συμβολή σου και η παρέμβασή σου για το μέλλον της Ευρώπης και όλοι έχουμε την αίσθηση ότι βλέπουμε πώς μιλάει η Ευρώπη, πώς μιλάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήταν καλό στο μέλλον να έχουμε πιο πολλούς πρωθυπουργού πρώην μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό πραγματικά το απολαύσαμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό πραγματικά που μου άρεσε είναι ότι ξεκινήσατε με αισιόδοξο μήνυμα Μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης, μιλάμε για τη χώρα σας, τη Λετωνία, μια επιτυχής ιστορία τις τελευταία χρόνια και με την υποστήριξη του κυρίου Ντομπρόφσκη υπό την ηγεσία του. Μεγάλη οικονομικέ επιτυχίε, μεγάλη επιτυχία για τη χώρα σε ό,τι αφορά τι επενδύσει τι οποίε ανέφερε ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και για το αίσθημα τη ασφάλεια, ότι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ασφαλεί και προστατευμένοι, γιατί αυτό είναι τμήμα μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά και τη Ρωσία και τι εξωτερικέ απειλέ. Είναι επιτυχημένη ιστορία γιατί μιλάμε για την ε, εντολή που μας έχει δοθεί. Αυτό το αναφέρε και ο κύριος Γιούγκα. Ανέφερε το τι επιτύχαμε στο θέμα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων εκατομμύρια νέων θέσεων απασχόλησης ε, που συστήθηκαν με το πρόγραμμα Γιούγκα, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κορονίδα ήταν ε, ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής. Άρα δηλαδή μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι για όλα αυτά που καταφέραμε από την καθοδήγηση του κυρίου Γιούγκα. Και κάτι άλλο. Εγώ με 46 ετών είμαι, ε, ανήκω σε αυτή την γενιά που μπορεί να πει ότι έζησε εν ειρήνη η προηγούμενη γενιά, ε, ναι, είχε και αυτή ειρήνη, αλλά είχαμε το σιδηρούν παραπέτασμα και η προπροηγούμενη γενιά είχε πόλεμο. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να το έχετε κατά νου όταν θα κάνετε την προεκλογική σας εκστρατεία. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα το να ζούμε στην Ευρώπη και θα προστατεύσουμε την Ευρώπη από όλους τους ε, εθνικιστές και τους εγωιστές. Το δεύτερο θέμα που αναφέρατε είναι εκείνο που είναι πολύ συγκεκριμένο, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, στις ανησυχίες των ανθρώπων. Αναφέρατε τη μετανάστευση. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που είπατε για την προστασία των συνόρων μας. Ε, ε, Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ένα ε, φιλόδοξο πρόγραμμα και χρειαζόμαστε και ένα πρόγραμμα για την Αφρική. Ίσως στο μέλλον να έχουμε και έναν επίτροπο για την Αφρική που θα συνδυάζει όλα αυτά που χρειαζόμαστε για την Ήπειρο αυτή. Ε, ξάλλου, τα περιφερειακά ταμεία είναι καθοριστική σημασία. Ε, το εμπόριο είναι καθοριστική σημασία και η κοινή αγορά. Πρέπει να ενισχυθεί η κοινή αγορά γιατί Καταρχήν, πρώτα απ' όλα πρέπει εδώ να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Και τέλος και η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά υπάρχουν στο θεματολόγιο, αλλά όταν μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. Γιατί υπάρχει ένα πράγμα που είναι απόλυτα σαφές, εντάξει είναι η πολιτική προσέγγιση, αλλά το άλλο σημαντικό θέμα είναι η μέθοδος. Πώς θα επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη Ευρώπη, αλλά υπάρχει το πρόβλημα της ομοφωνίας. Εγώ το αποκαλώ πρόβλημα την ομοφωνία. Γιατί ας πούμε όταν πρόκειται για τη Ρωσία πρέπει και 27 χώρες να συμφωνήσουν. Γι' αυτό πρέπει να αρθεί η ομοφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ένας ισχυρός πολιτικός παίκτη ε, με παγκόσμια και ουσιαστική εμβέλεια. Άρα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγέ. Και όταν μιλάμε για μεθόδους ε, νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή τη μέθοδο της ε, έγερση γεφυρών. Ας αναφερθούμε στη δική μου τη χώρα, η Γερμανία. Η Γερμανία ήταν ε, κατά της άποψης ε, του να υπάρχουν συγκεκριμένες ποσοστώσεις ε, για την κατανομή των μεταναστών μέχρι το 2015. Το 2015 ναι, γιατί, γιατί τότε εμφανίστηκε το πρόγραμμα στη Γερμανία και μέσα σε τρεις μόνο μήνες η Γερμανία άλλαξε γνώμη και ζήτησε ένα δεσμευτικό μηχανισμό ποσοστώσεων στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει κανείς να εξετάζει τα προβλήματα της Ευρώπης κάτω από εγωιστικό πρίσμα. Πρέπει να μάθουμε να έχουμε κατά νου και τη θέση των υπολείπων και των άλλων όταν, εάν μάλλον θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη. Και τέλος ένα μήνυμα, ε, μια Ευρώπη δημοκρατική. Γνωρίζετε για τι πράγμα μιλάμε. Είναι θέμα δικαιώματος ανάληψης ε, πρωτοβουλία. Το να μπορεί το Κοινοβούλιο να διεξάγει περισσότερες έρευνες, να εξετάζει και το Κοινοβούλιο την εφαρμογή των κανόνων και χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Πρωθυπουργέ που στηρίζει στην ιδέα του Spitzenkandidat, του βασικού εκπροσώπου μια ε, πολιτική ομάδα. Εγώ, παραδείγματο, χάρη, είμαι Spitzenkandidat και ε, ζητώ την υποστήριξή σα. Και τέλο μέλλον τη Ευρώπη σημαίνει ότι πρέπει να προστατεύσουμε την πεμπτουσία τη Ευρώπη. Μιλήσαμε για δημοκρατικό τρόπο ζωή, αλλά δημοκρατία ανεξάρτητη από τη δικαιοσύνη, ίση μεταχείριση όλων των ανθρώπων και δικαίωμα στην ελευθερία έκφραση, στην ελευθερία του τύπου, όλα αυτά τα δικαιώματα πρέπει να τα εγγυηθούμε στο μέλλον να υπάρχει ο απαραίτητος μηχανισμός. Να δώσουμε στον κόσμο ε, το καλό πρότυπο, το καλό παράδειγμα, πώς μπορεί κανείς ε, να ζει σε μια δημοκρατική Ευρώπη με ανθρώπινο τρόπο. Ο δημοκρατικός τρόπος ζωής είναι μια προσφορά στην Ευρώπη και αυτό ακριβώς είναι το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και... τώρα για τους σοσιαλιστές, η κυρία Μπρέσο παρακαλώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη τιμή σήμερα να σας καλωσορίσω, καθώς έχετε αναλάβει τα νέα σας καθήκοντα ω Πρωθυπουργό σε αυτό το ημικύκλιο. Και εσείς φυσικά το γνωρίζετε καλά, γιατί ήσασταν Ευρωβουλευτή περίπου για 10 χρόνια και είναι ακόμα μεγαλύτερη τιμή γιατί εσείς είχε, είστε όχι μόνο ο τελευταίος αρχηγός κυβέρνησης πριν από τις επόμενες ευρωεκλογέ, αλλά επειδή στην ομιλία σας αναφέρατε σημαντικές προοπτικές για την Ένωση που θα έχουμε το καθήκον να οικοδομήσουμε μετά τις 26 Μαΐου. Και γι' αυτό τον λόγο σας καλωσορίζουμε εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ως τελευταίος αρχηγός κυβέρνησης που έρχεστε να επισκεφτείτε το Κοινοβούλιο με τι εκλογέ. Η επίσκεψη σας αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για να συζητήσουμε για τη χώρα σας, τη Λετωνία και το ρόλο τη εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μα, ε, τους ευρωβουλευτές, είναι πάντοτε κάτι θετικό να συναντάμε έναν από τους ε, πρώην συναδέλφους μα ε, να εκπροσωπούν μια εθνική κυβέρνηση και ελπίζουμε να αυξηθούν οι συνάδελφοι. Εδώ ε, θέλουμε να εκφράσουμε μια συγκεκριμένη φιλοδοξία των Ευρωπαίων πολιτών, να οικοδομήσουμε μαζί μια ισχυρή ένωση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του καιρού μας. Ε, μένει μόνο ένα κράτος μέλος, ε, είτε πρόκειται για ένα μικρό κράτος όπως το δικό σας, είτε για μια μεγαλύτερη χώρα όπως η Ιταλία ή η Γαλλία. Ε, μπορεί κανένας να κάνει μόνος του τίποτα για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή, ούτε να ε, διασφαλίσει τη δική του άμυνα ή την οικονομική ανάπτυξη της χώρας του. Κύριε Γιούνκερ, όπως και εσείς και εγώ ε, αγαπώ την Ευρώπη, αλλά αγωνίζομαι για τα ενωμένα ευρωπαϊκά κράτη, στον πληθυντικό. Και επομένως ε, δεν βλέπω που είναι το πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάντως για τη δεσμευσή σας για την Ευρώπη και από την πλευρά της δικής μας ομάδας ε, καθώς ε, είναι η τελευταία παρουσία σας στο Κοινοβούλιο σήμερα, όπως είπατε. Εμείς ε, έχουμε εκτιμήσει τη δέσμευσή σας για μια Ενωμένη Ευρώπη που ίσως να πηγαίνει πιο πέρα από τα Ενωμένα κράτη της ε, Ευρώπης. Ελπίζουμε όσα είπατε να αποτελούν μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δέσμευση της κυβερνήσής σας, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, που μέχρι τώρα έχει δείξει κάποια αμφίσιμα σημεία σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊστικό σας χρώμα σε ένα πλαίσιο όπου τα μεμονωμένα κράτη δεν μπορούν να παίξουν ρόλο στη διεθνή σκηνή θα, μήπως ε, θα έπρεπε να θέσουμε τέλος τον κανόνα ομοφωνίας ε, στο Συμβούλιο που κι εσείς υποστηρίζετε. Ο κανόνας αυτός προωθεί μόνο τα μεμονωμένα συμφέροντα των κρατών μελών εις βάρος του γενικού συμφέροντος της Ένωσης. Θέλετε να συνεχίσετε να ε, αποτελείτε το φύλακα ενός κονκλαβίου όπου οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ή συχνά αναβάλλονται η παρουσία μιας ισχυρής Ευρώπης είναι κάτι απαραίτητο και το υπενθυμίσατε. Ε, θα πρέπει να δείτε που θέλετε να βρεθείτε στα βιβλία της ιστορίας από την πλευρά του συμφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών ή στην πλευρά όσων έχουν υποστηρίξει το συμφέρον ε, κάποιων ε, ελίτ και θέλω να επιμείνω. Θέλετε να βρεθείτε στην πλευρά όποιων ε, κατέστησαν ένα ε, ε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ή από την πλευρά σας όσους έδωσαν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα τα χρήσιμα εργαλεία προκειμένου να αναπτύξει τη δυναμική του. Για μας, για του σοσιαλιστές και δημοκράτες, η Ευρώπη οικοδομείται μέσω του νόμου και με σεβασμό φυσικά, ε, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, αλλά και των δικαιωμάτων των πολιτών. Από τον Ιανουάριο ε, κάποιες δηλώσεις που κάνετε έχουν προκαλέσει πολλές ερωτήσεις και θέλουμε απαντήσεις σε σχέση με την ευρωπαϊκή δέσμευση για την κατάσταση των προσφύγων στην Ευρώπη. Εσείς είπατε ότι είστε κατά. Όμως, πώς ε, θα γίνει αυτή η ανακατανομή ε, όταν ε, έχουμε κοινά σύνορα. Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ελεγγύης που εφαρμόζεται σε όλες τις κοινοτικές μας πολιτικές, παραδείγματος χάρη και στην πολιτική συνοχής. Τι μπορείτε να μας πείτε λοιπόν συγκεκριμένα για αυτό το ζήτημα. Τώρα, τι λέτε για την έρνησή σας να υποστηρίξετε την έρεξη σε υπερβάσιμα του άρθρου 7 κατά Πολωνίας και Ουγγαρία. Πώς εξηγείτε αυτή την έρνησή σας με τις σωστές επικρίσεις στην πολιτική του Πούτιν και την υποστήριξή σας σε κάποια μέρη ε, της ε, ε, δεξιάς από το Σολβίνι στον Όρμπαν τώρα. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι αυτό αποτελεί αντίφαση και τελευταίο σημείο, αλλά σημαντικό ποια είναι τα μέτρα που έθεσε εφαρμογή η κυβέρνησή σας σε σχέση με την όξυνση των διακρίσεων απέναντι στους ΛΟΑΔΜΑ στο ε, στην Ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού, αυτή η Επιτροπή δείχνει πολύ μεγάλες δυσλειτουργίε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση μέτρων για την προστασία των μειονοτήτων. Η Ένωση μας προωθεί ε, την ε, ανοχή και ε, εσείς θα πρέπει να σέβεστε τις αξίε. σα. ευχαριστώ Κνέου, νέου για την ομιλία σας και για τις απαντήσεις που θα δώσετε Στι ερωτήσει μου. Ευχαριστώ. Τώρα το ρόλο έχει ο κύριο Τσίλα από το ECR. Πρόεδρε, Χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Πρωθυπουργέ που σας έχουμε εδώ και που άκουσα το τόσο όμορφο περιεχόμενο της ομιλίας σας. Θα ήταν πολύ καλό να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Θέλω τώρα να επιστήσω την προσοχή σας και στις κυρίες που συνοδεύουν τον ε, κύριο Κάρινς. Μπορούμε να είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτές. Είναι γυναίκες της διπλωματίας και πράγματι είμαστε περήφανες για αυτές. Θυμάμαι την ημέρα που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Πολλές φορές όμως έχω λυπηθεί για διάφορες πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως επίσης και για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι τόσο καλή. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να μιλήσω. Η ομιλία σας δεν είπε ότι όλα είναι ωραία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ας συνεχίσουμε ειρηνικά να εκτιμούμε τα επιτεύγματά μας και να φροντίσουμε για μια ακόμα πιο ενωμένη Ευρώπη. Χαίρομαι που βάλατε αποχρώσεις αυτό. Το ECR ήταν πάντα η πολιτική οικογένεια η οποία υποστήριζε την πραγματική ενιαία αγορά σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Και ξέρω ότι έχετε κι εσείς κάποιες αμφιβολίες. Είπατε ότι δεν χαίρεστε πάρα πολύ με τους Ευρωπαίους ε, πρωταθλητές. Οι εθνικοί πρωταθλητές ίσως να είναι κάτι καλύτερο. Έχουμε διαφωνήσει και με τον κύριο Βέμπερ που λέει ότι θέλει να αλλάξει κάποιες αρχές που διέπουν τις κρατικές επιχορηγήσεις. Νομίζω ότι είναι ένα λάθος μήνυμα προς την οικονομία. Γιατί ωραία, ωραίο το μήνυμα η Ευρώπη που προστατεύει, αλλά που προστατεύει από ποιον, από τον έξω κόσμο. Εντάξει, αλλά τελικά μήπω είναι αυτό ο λάθο δρόμο, μήπω οι περισσότεροι κίνδυνοι υπάρχουν μέσα στην εσωτερική αγορά. Και εδώ μπορώ να σα δώσω παράδειγμα, στο οποίο αναφερθήκατε λίγο πολύ κι εσεί, που είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε για τα μηδενικά τέλη με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Πρόσφατα εγκρίναμε το πακέτο κινητικότητας. Πολύ επίμαχο θέμα. Και είναι σαφές ότι πολύ ωραία πολλές κυβερνήσεις βαλτικές και από διάφορες πολιτικές οικογένειες ήταν κατά. Οπότε τελικά είναι να αναρωτιόμαστε αν είναι κάτι κακό για τις χώρες της Ευρώπης, είναι δυνατόν να είναι καλό για την Ευρώπη την ίδια. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε το ίδιο πακέτο κινητικότητας ε, για τις εμπορικές μεταφορές στις Ηνωμένε Πολιτείε, ώστε να μπορεί κανείς με τον ίδιο τρόπο να κυκλοφορεί από τη Νέα Υόρκη στο Wyoming, θα ήταν καταστροφικό αυτό. Εμείς εδώ μιλάμε για το 1% του ΑΕΠ και ξεχνάμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο είναι το 20% του Αμερικανικού ΑΕΠ. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα πούμε. Και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια περισσότερη φεντεριλιστική Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν θέλει βέβαια το ΙΣΙΑ, το θέλουν άλλες πολιτικές ομάδες. Έχει καταφέρει πολλά η Λετωνία στην νομοθεσία της για τους μετόχους, για παράδειγμα. Στο Tax 3 δεν αναφέρθηκε όμως. Και δεν αναφέρονται ε, σαν κακά παραδείγματα άλλες ε, χώρες που δεν βρίσκονται και πολύ μακριά από εδώ από το Στρασβούργο. Έπειτα η έρευνα και η τεχνολογία φυσικά και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και φαίνεται αυτό από το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Εσείς το είπατε, αλλά πώς γίνεται η κατανομή. Δημογραφικά θα συνεχίσουμε ακόμα και με ένα ευρύτερο πρόγραμμα, το Horizon α πούμε που είναι ένα καλό πρόγραμμα, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τις δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη που οι διαφορές οι δημογραφικές θα ενισχυθούν στο μέλλον. Αλλιώς θα είναι το δημογραφικό στις περιφερειακές χώρες όπου θα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και αλλιώς θα είναι η κατάσταση στο κέντρο ή στο νότο. Θα υπάρξουν διαφορές ακόμα μεγαλύτερες από ό,τι έχουμε τώρα. Οπότε σε πολλά συμφωνώ μαζί σας, σε πολλά θέλω να πάω ακόμα πιο μακριά. Ελπίζω το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μια δικιά μας μεγάλη πολιτική οικογένεια ώστε να μπορέσει να ενισχύσει την ενή αγορά που είναι και βασικά ο πυρήνας της Ευρώπης και που θέλουμε να αναπτυχθεί περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστούμε εκ μέρους των φιλελεύθερων ο κύριος Στελίτσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρωθυπουργέ, λοιπόν, ε, καλωσορίσατε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Στην αρχή της ομιλίας σας κάνατε ένα σχόλιο ότι μάθατε πάρα πολλά πράγματα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Άρα και εγώ ε, θα κάνω ένα παραλυσμό, ένα ψεύτικο θα έλεγα, γιατί με βάση αυτή την παραδοχή θα ήθελα ο Τσέχος ε, Πρωθυπουργό ε, να είναι μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τότε θα είχαμε μια τελείως διαφορετική πολιτική της τσεχικής κυβέρνησης για τα ευρωπαϊκά θέματα. Αλλά πέρα από αυτό έχετε ένα πλεονέκτημα. Έχετε γνώση και σωστή τοποθέτηση. Νομίζω ότι αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία, αλλιώς δεν μπορεί κανείς να εξελιχθεί. Φοβάμαι όμως ότι όλα αυτά δεν συμβαδίζουν με τον παραλυσμό που έκανα με τον Τσέχο. Πρωθυπουργό. Αναφέρατε επίση το θέμα των γλωσσών. Είμαι σίγουρο ότι μιλάτε πολλέ γλώσσε ή τουλάχιστον καταλαβαίνετε πολλέ γλώσσε. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνετε τσέχικα, αλλά θέλω να σας πω, αυτά που είπατε είναι σαν να διαβάζει κανεί το εκλογικό μανιφέστο του δικού μου του πολιτικού κινήματος και αυτό βέβαια καλό είναι, θετικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το γεγονό ότι ανήκετε στο ΕΛΚ, εγώ ανήκω στου φιλελεύθερου, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα επί των οποίων μπορούμε και πρέπει να αναζητήσουμε ευρωπαϊκέ λύσει. Μία σειρά θεμάτων επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε και με άλλα κόμματα και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να στοχεύουμε στι επικείμενε εκλογέ. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά θέματα επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε και θα επιλέξω κάποια θέματα που θίξατε. Απλουστευμένε ε, λύσεις. Αναφερθήκατε σε εθνικιστές, σε λαϊκιστές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τα αίτια αυτού του προβλήματος. Τα αίτια των ανησυχιών και της ανησυχίες εκείνων που κάπου τους χάσαμε σε αυτή τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Αλλά πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς και δίκαιοι και να πούμε ότι έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Ότι και στις δικές μας τις πολιτικές οικογένειες, στις δικές μας τις πολιτικές ομάδες και τα κόμματα βρίσκουμε εκείνους που προσφέρουν τις απλουστευμένες ή υπεραπλουστευμένες λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ε, δούμε τι ακριβώς γίνεται στο πολιτικό τοπίο. Όσον αφορά άλλα θέματα που θίξατε, μιλήσατε για την εσωτερική αγορά, την κοινή αγορά. Νομίζω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο δεν υπάρχει κανείς που να μην πιστεύει ότι η εσωτερική αγορά ε, δεν έχει ε, να παρουσιάσει επιτυχίες, ότι πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω. Πράγματι, μόνο το 35% της εσωτερικής αγοράς είναι ανοιχτό, άρα δηλαδή υπολείπεται ένα 65%. Ε, επίσης, είπατε με απόλυτη σαφήνεια ότι υπάρχει συγκεκριμένο λόγο ε, να ε, πηγαίνει κανεί στι ΗΠΑ να κάνει δουλειέ, γιατί εκεί στι ΗΠΑ ε, είναι μια ανοιχτή αγορά. Στις ΗΠΑ μία έγκριση και αδειοδότηση χρειάζεται κανεί. εδώ, εδώ 28. Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι ότι αν πραγματικά θέλουμε μία σωστή εσωτερική αγορά, πρέπει να έχουμε μία ρυθμιστική αρχή για μία ενωμένη αγορά. Επίσης, ε, κάνατε παραλυσμό με τον αθέμητο ανταγωνισμό από την Κίνα και από αλλού. Και συμφωνώ πάλι μαζί σας, δεν πρέπει να επιβάλλουμε προστατευτισμό, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν ανοίξουμε τις αγορές, και εγώ με πέρα αυτού, τότε το πλεονέκτημα θα είναι στην πλευρά εκείνων που απατούν και εκείνων που είναι μεγάλοι. Γι' αυτό λοιπόν να μην έχουμε αυταπάτε. Θα έχουμε εσωτερική αγορά και ξαφνικά οι νεοσύστατε επιχειρήσει ε, θα είναι στην διαθέση όπω η Microsoft. Άρα δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε στα πρότυπα, στι προδιαγραφέ, στην πολιτική ανταγωνισμού. Άρα δηλαδή να έχουμε ένα θεμητό πλαίσιο και το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο να έχουμε το θάρρο και τη βούληση να συστήσουμε μια αμυγό εσωτερική αγορά κατά 100%, όχι μόνο 35%. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Επίσης, μιλήσατε για το θέμα των εξωτερικών συνόρων. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, είναι καθοριστική σημασία στο θέμα, αλλά εκεί εξακολουθούμε να αποτυγχάνουμε. Φοβάμαι λοιπόν, αν δούμε λιγάκι την Τσεχία, εκεί υπάρχουν ε, πολλοί ε, που διστάζουν, δεν έχουν τη βούληση να κατανοήσουν ότι ε, όταν θα έχουμε εσωτερική αγορά και ελεύθερη μετακίνηση, τότε πραγματικά θα μπορούμε να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας. Τέλος, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και πάλι, ως προς την κλιματική αλλαγή θα μπορούσαμε να δουλέψουμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα και το τελευταίο σημείο ε, θίξατε την κοινή γεωργική πολιτική, την σωστή μεταχείριση των αγροτών. Πράγματι, δεν έχουμε κοινή γεωργική πολιτική γιατί ε, σε πάρα πολλούς εθνικούς ε, προϋπολογισμούς ε, προβλέπονται επιπρόσθετες επιδοτήσεις πέρα από τις προβλεπόμενες. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση των επιχειρηματιών, των καταναλωτών και βεβαίως και των γεωργών. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει, λέει ο Πρόεδρος, να σεβόμαστε το ο χρόνο που έχει προβλεφθεί για τον κάθε ένα από εσά, έτσι ώστε να υπάρχει και χρόνο για τη διαδικασία Catch the Eye. Εκ μέρους της Ενωμένη ο κύριο Παπαντιμούλη. Η σημερινή συζήτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί σε λίγες ώρες ολοκληρώνονται οι εργασίες της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι η τελευταία ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ ενώπιον της Ολομέλειας και υποδεχόμαστε τον λετονό πρωθυπουργό ο οποίος ήταν και για εννιά χρόνια συνάδελφός μας στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και είναι ο δωδέκατος πρωθυπουργός που έρχεται εδώ να συζητήσουμε για το μέλλον της ευρώπης σαράντα μέρες πριν τις σημαντικές ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας. δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να αυτοεπαινούμαστε και να επισημαίνουμε τα κάποια θετικά που έχουν γίνει αλλά να δούμε το μέλλον τις προκλήσεις του μέλλοντος και όσα δεν έχουμε κάνει ή όσα έχουμε κάνει λάθος για να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε την ανερχόμενη λαϊκίστικη ακροδεξιά που θέλει να διαλύσει και την ευρωπαϊκή ενοποίηση ως σχέδιο και να διαλύσει τις κοινωνίες μας αναφερθήκατε κύριε κάρινς στον μύθο τον αρχαιοελληνικό του εσώπου με τις βέργες. μία βέργα σπάει εύκολα πολλές βέργες μαζί δεν σπάνε. σωστό. αλλά πρέπει να δούμε εμείς στην ευρωπαϊκή ένωση πού βρισκόμαστε δέκα χρόνια μετά την κρίση της lehman brothers. έχουν μεγαλώσει οι ανισότητες οι κοινωνικές και οι περιφερειακές έχει υποχωρήσει μέσα στην ευρώπη το κράτος δικαίου και η κοινοβουλευτική δημοκρατία το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και η κομισιόν έχουν ζητήσει εναντίον των κυβερνήσεων της πολωνίας και της ουγγαρίας την ενεργοποίηση του άρθρου 7 και στο συμβούλιο δεν κάνετε τίποτα απέναντι στις παραβιάσεις της δημοκρατίας το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και η κομισιόν έχουν ολοκληρώσει μια πρόταση για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών ασύλου επτά συνολικά φακέλους και στο συμβούλιο οι κυβερνήσεις δεν κάνετε τίποτα. η κομισιόν η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και το ευρωκοινοβούλιο θέλουν την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης με τον τρίτο πυλώνα που αφορά στο ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων και στο συμβούλιο δεν κάνετε τίποτα. ακριβέστερα κάποιες κυβερνήσεις όπως της γερμανίας και της ολλανδίας ουσιαστικά έχουν βάλει βέτο. αν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσει η ευρώπη και να γίνει πιο ισχυρή η πολιτική ενοποίηση ισχυρότερη η πολιτική διαφάνεια να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όπως μας ζήτησε χθες η 16χρονη γκρέτα τούνμπεργκ τότε θα πρέπει να σταματήσει η ευρωπαϊκή ένωση κύριε βέμπερ να είναι μια ομάδα κρατών όπου συζητούν 28 και στο τέλος αποφασίζουν οι γερμανοί. αυτό πρέπει να αλλάξει. και θέλω να σημειώσω ότι συμφωνώ με την παρατήρηση του προέδρου Γιούνκερ, ότι για να υπηρετήσουμε τους στόχους που έχουν τεθεί χρειάζεται και ένας ισχυρότερος κοινοτικό προϋπολογισμός με περισσότερα χρήματα στο κοινό ταμείο γιατί πρέπει να μην περικοπούν αλλά αντίθετα να ενισχυθούν τα κονδύλια για την κοινωνική συνοχή. Να μην περικοπούν, αλλά αντίθετα να ενισχυθούν τα κονδύλια για την κοινή αγροτική πολιτική να δώσουμε περισσότερα χρήματα για την νεολαία το erasmus την απασχόληση την έρευνα την καινοτομία και σας ρωτώ κύριε Κάνης, ως εκπρόσωπο του συμβουλίου αλλά και ως παλιό ευρωβουλευτή γιατί έχετε πετάξει στα σκουπίδια τις προτάσεις της επιτροπής μόντι για την αύξηση των ιδίων πόρων. πώς μπορεί να προχωρήσει η πολιτική ενοποίηση της ευρώπης η οικονομική ολοκλήρωση της ονε η νομισματική ενοποίηση χωρίς να κοιτάμε το κοινωνικό θέμα. Κύριε Γιούνκερ και κύριε Κάριν, στο Γκέτεμπορκ εγκρίθηκε η κοινωνική ατζέντα, αλλά παραμένει μια απλή ετικέτα. Δεν έχει αποκτήσει περιεχόμενο. Και όσο αυξάνονται οι ανισότητες, θα κερδίζει έδαφος ο λαϊκισμός των ακροδεξιών που θέλουν να διαλύσουν και την Ευρώπη και τη δημοκρατία. Πριν 80 χρόνια οι πολιτικοί πρόγονοι του κυρίου Σαλβίνη, της κυρίας Λεπέν, του κυρίου Όρμπαν, που κακώς τον κρατάτε κύριε Βέμπερ με αναστολή στις γραμμές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οδήγησαν στο φασισμό και τον ναζισμό και σε ένα πολύ νεκροπόλεμο. Αν θέλουμε λοιπόν να υπερασπίσουμε τη δημοκρατία, πρέπει στις επόμενες ευρωεκλογές να αποκτήσει μια ισχυρή πλειοψηφία μέσα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο η άποψη που λέει ότι χρειαζόμαστε μια περισσότερο ενωμένη πολιτικά δημοκρατική και κοινωνική ευρώπη που να μειώνει τις ανισότητες και να μην τις αυξάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάμπερτς από την ομάδα των Πρασίνων. Καλώ ήλθατε επίση στο Κοινοβούλιο, το οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά. Πάντοτε δεν συμφωνούσαμε στι οικονομικέ υποθέσει, αλλά πάντοτε ήμουν πολύ εντυπωσιασμένο από τη δέσμευσή σα για το κοινοευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και σήμερα είδαμε μια σχετική μαρτυρία. Και ε, πραγματικά ε, είναι τυπική η δέσμευση αυτή που βρίσκουμε στι δημοκρατίε τη Βαλτική. Πιστεύω ότι οι χώρε του Μπενελούξ με τι τρει χώρε τη Βαλτική θα πρέπει να συνεργαστούν βαθύτερα. Γιατί αν μπορούν να βρουν συμφωνίε μεταξύ του, νομίζω ότι θα μπορούσαν να οικοδομήσουν γέφυρε και να προωθήσουν την ενότητα στην Ευρώπη, ίσω καλύτερα από το γαλλογερμανικό ντουέτο που φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι κάπω τσακωμένο. Μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία σα μου άρεσε που μας υπενθυμίσατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ε, ένα project ειρήνης ε, και χρησιμοποιεί περισσότερο το διάλογο παρά τη βία. Αυτό είναι αιτιολόγηση όχι τον περασμένο αιώνα, αλλά η σημερινή αιτιολόγηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και μου άρεσε και η μεταφορά με το δεμάτι. Όπως και εσείς έρχομαι από μικρή χώρα, αλλά και μεγάλες ε, χώρες και μου άρεσε αυτό που είπατε για την ενιαία αγορά. Η ενιαία αγορά είναι η έσχατη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, γιατί παρόλο ε, που έχουμε τέτοιες συμφωνίες, διέπονται από τους δημοκρατικούς θεσμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλού δεν το βρίσκεται σε άλλε συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών. Επίση, μου άρεσε ε, το θέμα τη ήταν κάθετο για την νομοποίηση παράνομων εσόδων. Και μα αρέσει να ακούμε αυτά τα λόγια, γιατί ξέρω ότι είστε ισχυρά δεσμευμένο για το θέμα αυτό. Επίση, ε, ε, θα ήθελα επίση να διαφωνήσω όχι απαραίτητα με όσα είπατε, αλλά με κάποιε δράσει και θέσει τη κυβέρνηση τη Λετωνία. Ε, Καταρχήν, για μας τους πρασίνους, ε, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα πρέπει να αποτελέσει τη μηχανή, να έχει την ηγετική θέση της οικονομικής μετάβασης στις κοινωνίες μας. Αν δεν μπορέσουμε να τις κάνουμε να ταιριάξουν με τα όρια που μας θέτει η φύση, ε, απειλείται η ύπαρξη της ίδιας ανθρωπότητας. Είναι επίσης θέμα ηγεσία. Αν εμείς η Ευρώπη δεν έχουμε ηγετική θέση σε αυτή τη μετάβαση, άλλοι θα το κάνουν. Και τότε εμείς ε, θα μείνουμε με το να αγοράζουμε τις δικές τους λύσεις παρά να δίνουμε τις δικές μας στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, Μία περίπτωση και το αναφέρεται είναι η γεωργία. Εκείνη η αγροτική πολιτική είναι ο μεγαλύτερο προπολογισμό τη Ένωση. Θα πρέπει ε, κάθε λεπτό του ευρώ ε, που δαπανάται σε αυτή να συνεισφέρει στην μεταμορφώση του γεωργικού μα μοντέλου, έτσι ώστε να μειώνονται οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, να αποκαθίσταται η ποιότητα του εδάφου και η βιοπικιλότητα. Η κοινή γεωργική πολιτική προωθεί ένα πρωτοεκτηριστικό μοντέλο που καταφέρετε ε, κατά αυτών των στόχο και η κυβέρνησή σα ε, το υποστηρίξει και θεωρείτε ότι είναι πολύ πράσινο για τα γούστα σα. Καταλαβαίνω ότι η χώρα σα και συμφωνώ θέλει το δικό τη μερίδιο τη ε, ΚΑΠ. Όμω είμαστε πεπισμένοι ότι ο καλύτερο τρόπο να επιτευχθεί αυτό ο στόχο είναι να αγωνιστείτε για μια πιο πράσινη κοινή γεωργική πολιτική που απομακρύνεται από αυτό το πρωτοκριστικό μοντέλο και τη βιομηχανική γεωργία. Η δεύτερη πτυχή έχει να κάνει με την ηθαγένεια. Αναφέρεται τι ευρωπαϊκέ αξίε και αν διαβάσετε το άρθρο 2, η πρώτη αξία που αναφέρεται εκεί είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν ε, μπορεί να διαιρεθεί. Αφορά ε, όλους τους ανθρώπους και σήμερα και στο μέλλον. Η ε, Λετωνία, καθώς ανήκει χωρίς να θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταλήξει στον να είναι σημαντικό μέρος Σοβιετικής Ένωσης ε, έχει καταλήξει να έχει πάρα πολλούς ε, πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως ε, δεν πρέπει να διατηρεί απάτριδες 10% του πληθυσμού. Επίσης πρέπει να κάνετε περισσότερα, να προωθείτε τα δικαιώματα των μενοτήτων και να καταπολεμείτε τις διακρίσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τις αναπηρίες, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Τρίτον, ορίζουμε και σήμερα καταφέρετε να το αποφύγετε αυτό ότι και οι τρει δημοκρατίε τη Βαλτική έχουν ε, αποφύγουν ε, την ταξική στάση που έχουμε δει στο θέμα του ασύλου και τη μετανάστευση. Πραγματικά εκτίμησα τα λόγια σα στο θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, πρόσφατα η κυβέρνησή σα ε, δήλωσε ότι είναι αντίθετη σε οποιοδήποτε δεσμευτικό ε, σχέδιο μετεγκατάσταση, το οποίο μόνο αυτό θα οργανώσει την Ευρωπαϊκή Ελληνική. Επίση, αρνήθηκε να υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΙΕ για τη μετανάστευση το οποίο απλώς ε, παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Και εγώ και εσείς γνωρίζουμε ότι δεν είναι νομικά δεσμευτικό και βασίζεται σε αξίες ε, για τον επιμερισμό της ευθύνης, ε, της μη εισαγωγή διακρίσεως και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγνωρίζει ότι μόνο μια συνεργατική προσέγγιση θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Θα πρέπει όμως η Λετωνία να υπογράψει το έγγραφο αυτό. Και καθώ πλησιάζουν οι ευρωεκλογέ, αυτή είναι η τελευταία συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη, σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βασιστείτε σε εμά για να υπερασπίσουμε ακούραστα την ε, πρώτη ε, προσπάθεια για να οικοδομήσουμε μία ε, διεθνική δημοκρατία. Επίσης, βασιστείτε σε εμά για να την κάνουμε να λειτουργήσει για όλους, θέτοντα. Ε, στο επίκεντρο την οικονομική αξιοπρέπεια παρά τα οικονομικά κέρδη. Μία πιο ελεύθερη, βιώσιμη και δημοκρατική Ευρώπη είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες ε, και εμείς θα ζητήσουμε τη δική τους εμπιστοσύνη ακριβώς για να παράξουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και εξ του EFDD, ε, παρακαλώ κύριο Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ Κάριντς, αξιότιμε αντιπαλέ μου, ο Σανκλώτ Γιούγκερ, πρώτα απ' όλα σας εύχομαι καλό Πάσχα για το Πάσχα που έρχεται και να σας πω και τα εξή. Όλο αυτό το επεισόδιο με την Παναγία των Παρισίων δείχνει τελικά πόσο λίγο μας ενδιαφέρει η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης η ενότητα στην Ευρώπη που βασίζεται στην ελληνική φιλοσοφία, στο ρωμαϊκό δίκαιο, τη χριστιανική πίστη και την δημοκρατία θα έλεγα. Τελικά μας οδήγησε στη συνθήκη της Λισαβόνας και διαγράφηκε εκεί οποιαδήποτε μνήα στην χριστιανική Ευρώπη. Κάτι το οποίο όμως είναι ξένο προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το σχέδιό της αυτό για ε, κοσμική Ευρώπη έχει απορρίψει ουσιαστικά την ίδια τη δικιά μας πολιτιστική κληρονομιά και μας οδήγησε έτσι σε πολιτιστική αδυναμία, κάτι το οποίο καταδικάζουν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι ένα τρομακτικό οικοδόμημα καλτ ο Ροβεσπιέρος το είχε πει επίσης και με κάθε σεβασμό είπατε ότι η Ρωσία κάποια σχέση έχει με το Brexit. Μα συγγνώμη κύριε, οι Βρετανοί το 1940 πολέμησαν τον αυταρχισμό και είναι σε θέση να αποφασίζουν από μόνοι τους για το τι θέλουν ή δεν θέλουν από την Ευρώπη. Και δεν θέλουν γραφειοκρατικό αυταρχισμό από την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αλήθεια ότι είναι ε, μοναδικό, γιατί θέλει να είναι κυρίαρχο και το δικό μας, το δικό μας κοινοβούλιο κυριαρχεί μία ελίτ η οποία για πάνω από 30 χρόνια ηγείται από αυτούς τους Eurocult εύκολα μπορούμε να πούμε ότι φεύγουμε, ακολουθούμε τους κανόνες του ΠΕ και τίποτα άλλο. Αλλά οι Eurocalls αποφάσισαν διαφορετικά και αποφάσισαν, όπως η Πρωθυπουργό μας, να οδηγήσει την χώρα μας σε τόσες περιπέτειες. Ακούμε πολλές ανοησίες για διάφορα backstop στην Ιρλανδία και ότι τελικά μας απειλεί η Ευρώπη. Και αυτή η ευρωλατρεία μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Η κυρία Μέη αδίκως έχει αναγκαστεί να οδηγηθεί σε μία εντελώς παράλογη συμφωνία. Γιατί για να αποφευθούν οι ευρωεκλογέ, γιατί δεν θέλετε βέβαια να γίνουν, γιατί αν γίνουν θα κερδίσει το κόμμα του κύριου Φάραντ. Και αλλιώ αν δεν γίνουν αυτές οι ευρωεκλογέ στον Ηνωμένο Βασίλειο, επόμενες γενικές εκλογές εκεί θα κερδιθούν από το κόμμα του Brexit του κύριου Φάραντ. Οπότε λοιπόν αυτή η ευρωλατρεία πρέπει να φύγει από το Westminster. Ο κύριος Μπαρνιέ δεν είναι εδώ, ε? Πολύ καλός διαπραγματευτής και το Βρετανικό Κοινοβούλιο, τη έκπληξή του, δεν θεωρεί ότι πρόκειται για μια επιτυχία και λέει ότι δεν τη θέλει αυτή τη συμφωνία. Όμως αυτή η ευρωολατρία είναι ακόμα πιο σημαντική για αυτούς που πιστεύουν σε αυτήν και θεωρούν πιο σημαντικό να συνεχιστεί το οικοδόμημα αυτό όπως πηγαίνει τώρα αντί να πετύχουν μια καλή συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ηγείται με συνένεση και όχι με να θέλουν να τιμωρούν τους δε εκείνες τις χώρες, εκείνα τα άτομα τα οποία δεν συμμερίζονται την ίδια ευρωλατρεία. Συνεπώς, κυρίως από τις κάτω χώρες, ο κύριος Λάμπερτ, πρέπει ναι, να μαθαίνουμε από την ιστορία πράγματι αυτοί που έχουν ελεύθερη σκέψη από τις κάτω χώρες πρέπει να είναι παράδειγμα για μας. Δεν πρέπει να σταματάμε τον κόσμο από το να σκέφτεται και να αποφασίζει για τον εαυτό του. Η... Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η ιερά εξέταση στην Ισπανία που οδήγησε. Αυτοί λοιπόν που σκέφτονται ελεύθερα σήμερα είναι αυτοί που εσείς ονομάζετε λαϊκιστές. Εγώ προσωπικά προτιμώ να είμαι λαϊκιστής παρά όχι μη λαϊκιστής όπως είσαστε εσείς. Αυτό που εσείς περιγράφετε ως λαϊκιστές πολύ σύντομα θα εκλεγούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα έρθουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα κυριαρχήσουν εδώ. Και θα αλλάξουν ριζικά την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα καταστραφεί αυτή. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι που πρέπει να έχετε στο νου σας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερη απειλή στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, όπως ήταν η Ιερά Εξέταση τον 16ο αιώνα, που δεν επέτρεπε τη δημοκρατία και την ελεύθερη σκέψη. Κύριε, ο, ο Πρωθυπουργός Κάρενς είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τη μετανάστευση και ότι πολλοί θέλουν να έρθουν σε μια σταθερή δημοκρατική ήπειρο. Ε, δεν τους κατηγορώ. Κι εγώ, αν ζούσα στον τρίτο κόσμο ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, ναι, κι εγώ θα ήθελα να έρθω εδώ. Ποιο μπορεί να κατηγορήσει αυτού του ανθρώπου. Ναι, αλλά αν αλλάξουν τα νούμερα και αλλάξουν την ε, ίδια τη δημοκρατική φύση της Ευρωπαϊκής Υπήρου, τότε δεν ξέρω ποιοι θα θέλουν να πρωτοφύγουν από εδώ. Θα είναι μια καταστροφή. Το άλλο, ναι, είναι πιο ανησυχητικό από τα θέματα της υπηρεσίας υγείας. Τώρα, η Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει μόνο αν κυβερνάται με συνένεση και όχι σε βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, Πρόεδρος, έχετε δίκιο ο κύριος Κόμπουρν ξεπέρασε το χρόνο που είχε προβλεφθεί για εκείνον, αλλά άφησα και άλλους να υπερβούν το χρόνο τους. Ε, δεν είναι ότι όποιον συμπαθώ του δίνω χρόνο και όποιον δεν συμπαθώ δεν του δίνω. Οι κανόνες είναι όλοι για ίδιους. Περνάμε λοιπόν στον επόμενο μιλητή, στον κύριο Μπέι. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ, η τρομερή πυρκαγιά που χτύπησε την Παναγία των Παρισίων ε, μα κάνει να συνειδητοποιήσουμε το πόσο το χαρακτήρα έχει η πολιτιστική μα κληρονομιά μα, να ε, ένα από τα πιο ωραία κοσμήματα του ευρωπαϊκού μα πολιτισμού καταστράφηκε από τι φλόγες και μαύρησε την καρδιά των Γάλλων και των Ευρωπαίων. Ευτυχώ ε, η αξιοσημείωτη δράση των πυροσβεστών επέτρεψε να σωθεί ένα μεγάλο μέρο του κτηρίου που θα μπορέσει να αποκατασταθεί και να ξαναβρει το μεγαλείο του και με τη χαρά μαθαίνουμε ότι οι θησαυροί τη των Βεναγιάς των Παρισίων ε, σώθηκαν ε, όπως τον Καθήνο Στεφάνη. Όμως όλο αυτό οδήγησε στο να ε, συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε την κληρονομιά μας, αλλά και πιο γενικά την κληρονομιά του ευρωπαϊκού και χριστιανικού πολιτισμού. Κύριε Πρωθυπουργέ, αναφερθήκατε προλίγο σε αυτό που αποκαλείται ευρωσκεπτικιστές και θεωρείτε ότι είναι αντίθετοι στην ίδια τη ιδέα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εδώ κάνετε 100% λάθος. Πιστεύουμε στην Ευρώπη, είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχει ευρωπαϊκός πολιτισμός, μια, ένας πολιτισμό πολιτισμός και υπάρχει μια τεράστια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Όμως αυτή η βούληση απαιτεί επίσης και διάβια πνεύματος. Και είπατε για τη μετανάστευση δεν έχω λύση, δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε για να εμποδίσουμε τη μετανάστευση. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορούμε να δράσουμε και το δείχνει καθημερινό ο Ματέο στην Ιταλία. Όμω υπάρχουν δύο επιλογέ ξεκάθαρα. Αφενό, ο κύριο Ευρωμοπούλο, ο Ευρωπαίο Επίτροπο, μα είπε ότι χρειαζόταν μετανάστευση για να καλύψουμε το δημογραφικό έλλειμμα και αφετέρου η θεραλέα κυβέρνηση στην Ιταλία αλλά και στην Ουγγαρία που θεσπίζουν μεγάλε κοινωνικέ φορολογικέ πολιτικέ που υποστηρίζουν την οικογένεια και την ευρωπαϊκή γεννητικότητα. Υπάρχουν λοιπόν δύο ώρα πράγματα εδώ που συγκρέονται μεταξύ αυτών που δέχονται και ενθαρρύνουν τη μετανάστευση και όσοι το αντίθετο θέλουν ε, να σταματήσει το μεταναστευτικό ρεύμα και να ενθαρρύνουν την ε, γεννητικότητα στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από κατάργηση κάθε προστασία ε, με την εσωτερική αγορά, τον θεμητό ανταγωνισμό, με του απεσπασμένου εργαζομένου ε, και στο εξωτερικό, πολλαπλασιάζοντα ε, τι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών και τη μείωση των δασμών. Σήμερα, οι ΕΠΑ και η προστατεύουν τον εαυτό του, μπορούν να προστατεύσουν με κάθε τρόπο την εσωτερική του αγορά και φυσικά έχουν επιθετική στάση στον υπόλοιπο κόσμο και χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο ως ένα χώρο που μπορούν να δράσουν ελεύθερα συνήθως ε, εις βάρος ε, της δικής μας οικονομίας και των εργαζομένων μας. Ορίστε και εδώ έρχονται ε, σε αντίθεση δύο οικονομικά οράματα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο ως ένα εντελώς ανοιχτό χώρο και ένα άλλο όραμα που να προστεύεται οικονομικά και εμπορικά σε ό,τι αφορά τη θεσμική οργάνωση. Η Ευρώπη θα πρέπει ε, να προωθήσει την δημοκρατία μπροστά στην ε, τεράστια εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, άκουσα τι είπε και ο κύριος Βέμπερ και ο Μανώλη Μακρόν. Μας είπαν ότι πρέπει να πάμε ακόμη πιο μακριά στο φεντεραλισμό και να καταργήσουμε τον κανόνα της ομοφωνίας. Επίσης μας ζητούν και να καταργηθεί και η δική η πλειοψηφία και τέλος και απλή πλειοψηφία για να καταλήξουμε σε μια εντελώς πιο αδιαφανή λειτουργία και πιο αυτα και εδώ έχουμε δύο αντιτιθέμενα ορώματα. η Ευρώπη τη συνεργασία και των εθνών ή η Ευρώπη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιτάχυνση προ το φεντεραλισμό. Ε, απέχουμε πέντε εβδομάδες από τις ευρωεκλογέ. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ε, φυσικά είναι στο σταυροδρόμι ε, και έχει την ικανότητα η Ευρώπη να δώσει μια ευκαιρία προκειμένου να λάμψουν τα έθνη μας στην παγκόσμια σκηνή. Όμως θα πρέπει να σπάσουμε το μεγάλο δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και να απομακρυνθούμε από τη τεχνοκρατική λογική. Η Ευρώπη θα προστατεύσει την οικονομία της ή θα γίνει ο εξυπηρέτηση των άλλων μεγάλων δυνάμεων. Η Ευρώπη θα θέσει τα έθνη και τους λαούς ε, στο κέντρο του προγραμματός της ή θα διαλυθεί, θα υπερασπίσει τον πολιτισμό της ή την ταυτότητά της ή θα εξαφανιστεί. Ο κύριος Γκόλνης από τους μία γεγραμμένους, παρακαλώ. Κύριε Πρωθυπουργέ και αγαπητέ τελευταίο συνάδελφε, μας μιλάτε για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Α πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν φαίνεται αυτό το μέλλον πολύ λαμπρό αν δεν αλλάξουμε προπτική. Τα 30 χρόνια που είμαι εδώ σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είδα να αναπτύσσεται μια στρεβλή δυναμική των πολιτικών ομάδων ε, που θυμίζει κακές στιγμές. Πρόκειται για τις αρχές που διακηρύσει χωρίς όμως να τηρεί και έτσι είναι σε βάρος των διαφόρων μειονοτήτων. Νομίζουμε ότι έχουμε εντολή για να κανονίζουμε τα πάντα, ακόμα και τη σεξουαλική ζωή των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα υπερκράτος παγκόσμιο που να έχει ένα σωρό περιορισμούς κανόνες, αλλά να είναι ανοιχτό σε ανταγωνισμό με χώρες που δεν έχουν τίποτα ή πάρα πολύ λίγα. Η δικιά σας χώρα απελευθερώθηκε από το ζυγό της ε, σοσιαλιστικής χώρας ε, στην οποία βρισκόσαστε. Δεν νομίζω ότι θέλετε να έρθετε εδώ για να βρεθείτε σε έναν άλλο ζυγό. Πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Η Ευρώπη πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές αξίες του πολιτισμού μας. Να υποδέχεται τη ζωή και όχι την άμβλωση τη μαζική. Να θέλει την οικογένεια και όχι να την καταπιέζει συστηματικά όπως επίσης τις ε, σεξουαλικές μειονότητες. Εμπόρια, ε, πορικά αγαθά. Δεν είναι απαραίτητα αυτό που προσφέρει την ευτυχία και την ευημερία. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ ελεύθερων εθνών με συγκεκριμένα προγράμματα, με νούμερα και σε συγκεκριμένους τομείς όπου ο πολίτης να μπορεί να μετρήσει και το κόστος αλλά και το ωφέλη. Η επανάσταση των λαών κατά εκείνων που θέλουν να τους περιορίσουν, όπου περιορίζουν την ταυτότητά τους, έχει ξεκινήσει. Και εδώ ακόμα καταφέραμε να ρίξουμε τα τείχη του ψεύδους που εμπόδιζαν τους πατριώτες από διάφορες χώρες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Σε αυτό λοιπόν το βελούδινο περιβάλλον υποκρισίας οι λαοί αρχίζουν να ανοίγουν τα μάτια τους. Έχουμε σπήρι, άλλοι θα μαζέψουν τη συγκομιδή και για να διατηρηθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μας πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Ζήτω η ελεύθερη λαή μέσα σε μια ανανεωμένη Ευρώπη των Εθνών. Πρόεδρος, ε, ήμουν ευέλικτος ε, στον πρώτο γύρο των παρεμβάσεων, αλλά επειδή στις 12.30 πρέπει να ψηφίσουμε και θέλουν να μιλήσουν όλοι εκείνοι ε, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία Catch the Eyes, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρείτε το χρόνο που σας έχει δοθεί, γιατί αλλιώς θα αποκλείσετε κάποιους από το να λάβουν το λόγο. Και επειδή αυτή είναι η τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να φύγουν όλοι από την ολομέλεια ικανοποιημένη, Συμπεριλαμβανομένου και του Λετωνού Πρωθυπουργού, του κυρίου Κάριντς. Έχετε το λόγο για να δώσετε τις απαντήσεις σε αυτό τον πρώτο γύρο των τοποθετήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη μου παρέμβαση ήταν λιγάκι μακρά. Αυτή η παρέμβασή μου θα είναι πάρα πολύ σύντομη. Υπάρχουν δύο τρόποι για να αντιμετωπίζει κανείς τις διαφορές απόψεων. Ο καλύτερος τρόπος είναι αυτό που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, συζήτηση, ακούει ένας την άποψη του άλλου, σέβεται τον άλλον και τελικά ε, γίνεται η ψηφοφορία και προχωράει κανείς παρακάτω. Και υπάρχει και ένας άλλος τρόπος ε, για να γίνονται τα πράγματα, κάτι που η δική μου χώρα το βίωσε για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν ήταν υπό την κατοχή της ε, Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή να μην έχει κανείς το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του, να μην λέει τίποτα, κάποιος άλλος λαμβάνει τις αποφάσεις και σε συμπαρασύρει ή σε αφήνει κατά μέρο καθώς προχωράει. Ε, νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές ποιο είναι ο καλύτερο τρόπος ανάμεσα στους δύο. Εγώ είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με όλους όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε μαζί. Αυτή είναι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι κατορθώσαμε να διατηρήσουμε ε, κυρίαρχες χώρες με ισχυρές ταυτότητες, με τη γλώσσα τους, με τον πολιτισμό τους η κάθε μία, με ιστορία που βέβαια συνδέεται μεταξύ των διαφόρων χωρών πολλές φορές και παράλληλα κατορθώσαμε να ανοίξουμε τις αγορές στο εμπόριο. Μπορέσαμε να συνδυάσουμε, να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας και να εκφράζουμε μια ισχυρή φωνή στον κόσμο. Για κάποιον που δεν ξέρει τι είναι η Σοβιετική Ένωση, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Μα απολύτως τίποτα. Εδώ έχουμε μία ένωση ελεύθερης πολιτικής βούλησης ε, τα κρατημέλη είναι ελεύθερα να συμμετέχουν οι πολίτες επίσης ελεύθεροι να συμμετέχουν και βλέπουμε ότι αν οι πολίτες αλλάξουν γνώμη κανείς δεν τους εμποδίζει. Είναι μια πραγματικά ελεύθερη ένωση, είναι ένα μοναδικό εγχείρημα στον κόσμο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια χώρα που βασίζεται προέκυψε από τη μετανάστευση. Οι αρχαίγονοι Αμερικανοί δεν είναι και τόσο συνηθισμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχουν πολλοί εξ αυτών. Αυτοί τους οποίους ε, αποκαλούμε Αμερικανούς ε, σε γενικές γραμμές έρχονται από την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία. Ε, αφήνουν κάτι πίσω τους και γίνονται κάτι καινούριο όλοι μαζί. Στην Ευρώπη όμως κανείς από εμά δεν είναι αναγκασμένος να μετακινηθεί. Μπορούμε να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας, την ταυτότητά μας και συνεργαζόμαστε σε πολιτικό και οικονομικό πεδίο για να εκφράσουμε τα κυρίαρχα συμφέροντά μας. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν παρετούμεθα από τίποτα, συνδυάζουμε τους πόρου μα και από το να είμαστε απομονωμένοι και μεμονωμένοι είμαστε πολύ πιο ισχυροί ως μια ενωμένη Ευρώπη. Ευχαριστούμε και εμείς ε, κύριε Πρωθυπουργέ για την σύντομη ομιλία σας. Ο πρώτος που έχει το λόγο στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ είναι ο κύριος Κέλαμ. Κύριε Πρόεδρε, και για μένα αυτή είναι η τελευταία μου παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα νομίζω όσον αφορά την ρωσική επιθετικότητα πρέπει να διερωτηθούμε τι μπορεί να γίνει ακόμα και τι πρέπει να ληφθεί υπόψη για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την απειλή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιμείνει στο να εξισωθούν τα ε, εγκλήματα των ε, κομμουνιστών με αυτά των Ναζί. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει. Εάν η ΚΑΓΚΕΜΠΕ της ε, Σοβιετικής Ένωσης ε, όπως και η Γκεστάπο του Χίτλερ είχε καταδικαστεί με τον ίδιο τρόπο ως δολοφονική οργάνωση, τότε και τα στελέχη της Γκεστάπο, της Γκεστάπο, της Καγκεμπέ, δηλαδή της Ρωσίας, δεν θα μπορούσαν ε, σήμερα να ηγούνται της Σοβιετικής Ένωσης. Το κράτος που υπάρχει σήμερα υπάρχει μόνο λόγω της ε, διαφθοράς, της ευρωπαϊκής διαφοράς, ε, κλάπησαν χρήματα και οι Ρώσοι τα ξέπλυναν σε δυτικές τράπεζες. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτές τις ροές χρημάτων, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει πλέον, δεν θα μπορεί να επιβιώσει ο κύριος Πούτιν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κέλα που για τόσα χρόνια ήταν υποδειγματικός βουλευτής και το έχω πει δημόσια για μένα πάντοτε αποτελούσατε παράδειγμα προς μίμηση. Τρέφω μεγάλη εκτίμηση και θαυμασμό για σας, ε, γιατί έχετε αγωνιστεί για την ελευθερία της ε, χώρας σας και για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη συνεισφορά στο Κοινοβούλιο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόπες Αγγιλάρη ο επόμενο ομιλητή. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Κύριε Πρωθυπουργέ. Πρόκειται για το τέλος της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να δείξουμε σεβασμό στο ομιλία σας υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, είναι καιρός να αποτιμήσουμε τις συζητήσεις που είχαμε με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Να χαιρετήσουμε το έργο του Προέδρου Γιούνκερ ο οποίος έδωσε υψηλής ποιότητας απαντήσεις. Όμως, θέλω να πω κάτι αφού άκουσα την ομιλία σας. Μιλήσατε ε, όχι για την καταπολέμηση του λαϊκισμού, αλλά δεν είναι ασυμβιβαστό να τον καταπολεμήσουμε όταν ακούμε τέτοιες ε, ανοησίες εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να απαντήσουμε. Δεύτερον, μιλήσατε για τη μετανάστευση. Ναι, πρέπει να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είπατε τίποτα για αλληλεγγύη. Και αυτό αποτελεί μια εντολή τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για αλληλεγγύη και τη ε, την διαχείριση των συνόρων, ε, τότε αυτά θα πρέπει να τη διασφαλίσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ Κάριν. Σταρμπάτη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ο Ζαν-Κλοντ Juncker είπε ότι πρέπει κανείς να αγαπάει την Ευρώπη. Δίκιο έχει, και εγώ την αγαπάω. Αλλά ακριβώ όταν αγαπάει κανείς την Ευρώπη πρέπει να κατανοεί και τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέω ότι δεν πρέπει να θυσιάσουμε τους λαούς μας στο πομό της Ευρώπης Κύριε Ντομπρόφσκι, ε, ε, ξέρετε ότι οι νέοι μας ε, φεύγουν. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην μεταναστεύουν. Κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς είπατε ότι ε, χρειαζόμαστε αγορές μη ρυθμισμένες και έχουμε δύο κεντρικές αγορές που είναι απόλυτα ρυθμισμένες και έχουμε τις ισοτιμίες και τα επιτόκια. Εάν λοιπόν είναι συνεδεμένες οι ισοτιμίες με τα επιτόκια, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να παρισφρήσουν άλλοι παράγοντες, γιατί αν δεν συμβεί αυτό, τότε υπάρχει ένας σκληρός μηχανισμός προσαρμογής στην αγορά. Εύχομαι λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο μέλλον, να μην λέει κανείς ε, ότι ε, πρέπει να θυσιάσουμε τους λαούς μας στο βωμό της Ευρώπης. Όχι. Το εργατικό δυναμικό πρέπει να υπάρχει εδώ στην Ευρώπη. Το να ε, μην φροντίζουμε τον ανταγωνισμό, αυτό είναι το πρόβλημα. Τα κράτη πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και αυτό είναι το καθήκον που πρέπει να επιτελέσετε στο μέλλον. Ο κύριος Μητροφάνο, τους παρακαλώ. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχικά Ήθελα να μιλήσω για την φυγή κεφάλων ε, που βιώνουμε στη χώρα μας, ε, τη Λετωνία. Εμείς ε, χάνουμε τους νέους ερευνητέ μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει να αντιδράσω σε ένα μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Γιατί ζήτησε από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσουν το καλό παράδειγμα τη ολοκλήρωση στη Λετωνία. Πρέπει να πω, δεν είναι μια ιστορία επιτυχία. Είναι μια ντροπιαστική ιστορία ε, που στρέφεται κατά τη εκπαίδευση των μειονοτήτων. Ε, μετά την ανεξαρτησία, το μεγαλύτερο μέρο των μειονοτήτων ε, υποστήριζαν ε, την ανεξαρτησία και την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης χώρας. Όμως ε, τώρα τα παιδιά μας, τα παιδιά των οικογενειών των μειονοτήτων δεν μπορούν να μορφώνονται στη μητρική τους γλώσσα. Παρακαλώ μην ακολουθήσετε αυτό το παράδειγμα, συνάδελφοι. Κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, για 2.000 χρόνια στην χώρα μου είχαμε αυτή την τρέλα για την Ευρώπη. Η δικιά μου η χώρα δεν είναι ευχαριστημένη με την Ευρώπη. Όταν έχεις σωθεί από τα πεδία των μαχών, εξακολουθείς και θέλεις, να πιστεύεις, θέλεις την ειρήνη. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό ήταν ένα πείμα ενός Ούγγρου ποιητή το 83 και εσείς ε, ακούσατε τα πρώτα και τα τελευταία λόγια του πείματος αυτού. Και αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Θεός να φυλάει και να προστατεύει τη χώρα μου και τη χριστιανική Ευρώπη. Αντίο σας. Ο κύριος Βέρ τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ της Λετωνίας, σας θαυμάζω πολύ. Όχι μόνο γιατί γίνατε Πρωθυπουργό, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έχετε αναλάβει αυτό το καθήκον. Ήσασταν και προβλεφτή τώρα είσαστε από ένα μικρό κόμμα, καταφέρατε όμως να πετύχετε πλειοψηφία και να ηγηθείτε επιτυχώς τη σημερινή κυβέρνηση στη Λετωνία. Πράγματι, αξίζετε γι' αυτό, γιατί είσαστε ειλικρινή, τίμιο και έχετε πάρα πολλέ ικανότητε. Είσαστε μια επιτυχής ιστορία. Αυτό είναι και η ιστορία της Λετωνίας. Βέβαια, τώρα η βασική ερώτηση. Ζείτε σε μια χώρα που βρίσκεται σε μετάβαση, όπω και η δικιά μου η Σλοβενία. Το θέμα του κράτου δικαίου είναι πάντα πολύ επίκαιρο. Ήμασταν μάρτυρε ε, των ε, διαφόρων ε, κομμάτων και παραδόσεων και επεισοδίων που παρακολουθούμε. Εγώ πιστεύω ότι και άλλες χώρες σε μετάβαση έχουν προβλήματα με την δικαστική εξουσία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, να έχει δηλαδή έναν μηχανισμό ώστε όταν υπάρχει πρόβλημα με το κράτος δικαίου σε χώρες μετάβασης να κάνουν κάτι. Ευχαριστώ, η κυρία Πιλάρντε Καστιγιώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που έχουμε μπροστά μας ε, τον Πρωθυπουργό, είναι ένας εξαιρετικός ε, συνάδελφος, αλλά ε, δεν είναι μόνο αυτό. Κύριε Κάρνης, θέλω να πω ότι αφήσατε το αποτύπωμά σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρομαι τότε που ήσασταν συντονιστής, που είχατε υπό την καθοδήγησή σας πολλά σημαντικά θέματα. Αυτό όμω που σήμερα είναι το πιο σημαντικό είναι ότι μας παρουσιάσατε ένα όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσατε για το παρελθόν, το παρόν και το πιο σημαντικό για το μέλλον. Και ε, σε αυτό τον δρόμο πολύ σωστά αναφέρατε και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η κοινή αγορά. Πιο συγκεκριμένα η ενιαία ψηφιακή αγορά. Αναφέρατε το που ακριβώς βρισκόμαστε και ξέρετε πολύ καλά ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο διστάζει. Δεν είναι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο δεν αναχαιτίζει τους φραγμούς. Τώρα εσείς έχετε μία ε, πλεονεκτική προνομιούχο θέση στο Συμβούλιο, έχετε έδρα, Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι έτσι μπορείτε να προχωρήσετε πολύ πιο γρήγορα και να άρετε τους φραγμούς. Σας εύχομαι καλή τύχη. Καμπούλα Νάτρη, επόμενη ομιλήτρια. Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή να γνωρίζω τον Πρωθυπουργό ως καλό συνάδελφο στην Επιτροπή Ήτρε τότε που εργαζόμασταν για μια ε, ψηφιακή ενωμένη Ευρώπη. Ε, πραγματικά και εγώ με πολύ χαρά εργάζομαι για αυτήν την Ευρώπη όπου θα είμαστε αρκετά θαραλέοι για να εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι μπορούμε μόνο από κοινού να, ε, παρουσιά, να επιτύχουμε πάνω από 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ε, άρα λοιπόν αυτό το 20% είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα λαϊκίστικα που αναφέρονται, κλείστε τα σύνορα ή ε, μην κάνετε εμπόριο με άλλες περιοχές, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πώς αυτό θα βοηθούσε τους Ευρωπαίους. Αλλά όταν μιλάμε και για την κλιματική αλλαγή και εκεί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι από κοινού μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις ε, απλές οικογένειες που θέλουν να έχουν αυτοκίνητο. Όμως η αυτοκινητοβιομηχανία προσφέρει νέα αυτοκίνητα με μικρότερες ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Μπορούμε λοιπόν να τα καταφέρουμε όλοι από κοινού. Ως εκ τούτου προσβλέπω στον απευθυντή Ευρώπη στους ε, πολίτες της και κατά διάρκεια της προεκλογικής εκστρατεία. Νομίζω όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι εμείς έχουμε δουλέψει για να μπορούμε μπορούν οι εργαζόμενοι να μετακινούνται και πέρα από τα σύνορα, δουλέψαμε για να υπάρχουν καλύτερε συνθήκε εμπορίου και εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Ντεσμέικερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάριν. Πολύ ισχυρή η ομιλία σας, πολύ δυνατή για τα δημοκρατικά έθνη. Ωραία. Small is beautiful. Και η Λετωνία είχε κυριαρχία από πολύ ισχυρού γείτονε για πάρα πολλά χρόνια και τώρα έχει καταφέρει να έχει μια τεράστια επιτυχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το βλέπει αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλα έθνη, η Σκοτία, η Καταλωνία, που είναι ε, δημοκρατικά και δημοκρατικά προσπαθούν να ανεξαρτοποιηθούν και όμως αυτό φαίνεται να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εδώ. Και εξού και η βία σε βάρος των ψηφοφόρων στην Καταλωνία από τους ηγέτες της Ισπανίας. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μόνο όταν δούμε ότι το δημοκρατικό δικαιώμα, τα δημοκρατικά δικαιώματα των λαών γίνονται σεβαστά. Και δεν μπορεί να μιλάμε χωρίς να κάνουμε αυτά που λέμε. Χοκμάρκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Οι εξελίξεις στην Λετωνία, την Εσθονία, τη Λιθουανία αποτελούν το θαύμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Καταπληκτικά επιτεύγματα. Ελευθερία. Πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησα στην Σουηδία να στηρίζω. Ε, πριν στήριζα την ανεξαρτησία της Εστονίας, της Λετωνίας, της Λεθονίας, θυμάμαι, με τις Σάντρα του και ένα σωρό άλλους. Αγωνιζόμασταν για την ανεξαρτησία στην Σοβιετική επικράτεια. Και τώρα ένας καλός μου φίλος, εδώ δίπλα μου κάθεται, και εσύ ναι, Ήτανε ευρωβουλευτής και τώρα είναι επικεφαλής της κυβέρνησης της ελεύθερης Λετωνίας. Αυτό είναι το θαύμα. Και θέλω να το πω σε όλους τους συναδέρφους εδώ, γιατί και για μένα αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία εδώ. Ωραία, θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα, να σας είχαμε εδώ Κριστιανής Καρίνης. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να πω, δεν χρειαζόμαστε τους Φάρατζης και, και τους Κόμπερνς εδώ πέρα που να μας λένε ότι είναι καλύτερα να μην έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτά που εσείς καταφέρατε είναι ακριβώς ένα τεράστιο επίτευγμα. Μας δείξατε, είσαστε το ζωντανό παράδειγμα το ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και τι ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε. Εσείς, οι χώρα σας, οι χώρες μας είναι το καλύτερο παράδειγμα της Ευρώπης και είμαστε περήφανοι εμείς οι Σουηδοί, γιατί είμαι από τη Σουηδία, που σας είχαμε και, τον, και σας έχουμε γειτονική χώρα. Ευχαριστώ, Γκούναρ, ε, για το έργο σου στο Κοινοβούλιο αυτό. Συνάδελφο Μπόγκοβιτς. Καλημέρα σας, αγαπητέ Χριστίανα. Είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση να σε ξαναβλέπω. Είχαμε περάσει πολύ καλές στιγμές ως συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία σου. Ο Σλοβαίνος Πρωθυπουργό ε, είχε ε, προσκληθεί να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως απέριψε την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ λοιπόν για την υπέροχη ομιλία σου που ολοκληρώνει αυτό το ε, επεισόδιο όταν έρχονται αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων να μιλήσουν για το μέλλον της Ευρώπης. Η χώρα σου είχε μια δύσκολη ιστορία αλλά και εσύ είχες πέρα μια ιστορία, προέρχεσαι από μετανάστες γονείς και θαυμάζω τώρα πόσο δεσμευμένος είσαι για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αφενός και πόσο αφοσιωμένος είσαι στην ελευθερία αφετέρου. Είπες ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και σε ό,τι αφορά στην αγορά εργασίας, στην οικονομία κτλ. Σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέλω να θέσω την εξή ε, ερώτηση. Οι καθαροί συνεισφέροντες στο Συμβούλιο κατανοούν ε, ε, την έννοια της ελληνικής που μπορεί να εκφραστεί μέσω της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής αξίζει για να ε, καταβάλουν το 1 το το 1,3 του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Εγώ ελπίζω όμως ότι θα γίνει η Ευρώπη καλύτερη στο μέλλον. Μπλάνκο Λόπε, παρακαλώ, που Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Τη διάρκεια αυτής της θητείας ε, μπορέσαμε να συνεργαστούμε και το λέω στην τελευταία μου παρέμβαση αυτό στο Κοινοβούλιο. Να συνεργαστούμε λοιπόν για να έχουμε μια ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πιο ανταγωνιστική, με λιγότερες εκπομπές άνθρακας μαζί και με τον Επίτροπο Κανιέτα για να συνεργαστούμε για να έχουμε μια νομοθεσία που να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι η μεγάλη απειλή κατά του πλανήτη έχοντας μια οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα ιδιαίτερα φιλόδοξη γιατί ξέρουμε ότι η ενέργεια που δεν καταναλώνεται είναι η πιο καθαρή. Να συνεργαστούμε για την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δίσδυση και σίγουρα μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών του άνθρακα σε τομείς που ρηπαίνουν όπως ε, είναι η θέρμανση, η ψήξη και οι μεταφορές. Να συνεργαστούμε για να μειώσουμε τις εκπομπές και για να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα καθολικό νομοθετικό πλαίσιο που να μας καθιστά ε, σε μια ηγετική θέση για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Η Ευρώπη έχει μέλλον να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όπως πράξαμε σε αυτή τη θητεία καταπλημώντας το είναι πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ για τη δική σας συνεισφορά. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρωθυπουργέ, σήμερα ακούσαμε επανειλημμένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο παρουσιάζουν ε, εντυπωσιακά νούμερα και αναφέρεται και παραδείγματα. Συνεργαστήκαμε για θέματα καταπολέμησης της ε, διαφθοράς, επίσης ε, για την αντιμετώπιση της, παράνομης, ε, της νομιμοποίησης από παράνομα έσοδα. Όσον αφορά αυτό το ξέπλυμα του χρήματος, δεν είναι μόνο τα χρήματα που έρχονται από εγκληματικέ δραστηριότητες, αλλά και τα χρήματα που διοχετεύονται στην τρομοκρατία, στην παράνομη διακίνηση ανθρώπινων όντων. Στο επόμενο λοιπόν ε, κοινοβούλιο θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να μιλήσω εκτενώς ε, για τα θέματα αυτά. Επόμενος ομιλητής, Βαϊτέρε, παρακαλώ, η κυρία Βαϊτέρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Πρωθυπουργέ. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον Πρωθυπουργό μας. Ε, η ομιλία σου ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, ανέφερες και πολλά επώδυνα θέματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Είμαι επίση ε, ιδιαίτερα υπερήφανο που κατόρθωσε να συστήσει κυβέρνηση στην Λετωνία και με νέε δυνάμει όταν ε, παλιά στελέχη φοβόντουσαν. Εσύ όμως τα κατάφερες, μπροστά μας ε, έχουμε πολλά και δύσκολα. Βεβαίως ε, πρέπει να περιορίσουμε τις δαπάνες μας, διότι δεχόμεθα πλέον λιγότερα κονδύλια από τα Ταμεία Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άμεσες ε, πληρωμές ε, είναι μικρότερες από ό,τι σε άλλες χώρες ε, και όσον αφορά την κοινωνία ακούσαμε ότι συνεχίζεται αυτή η πολιτική ρωσοποίησης και εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε κατά αυτής. Αναφέρθηκαν και τα θέματα μειονοτήτων. Η Λετωνία είναι η μόνη χώρα όπου εξακολουθούμε να προσφέρουμε μια πλήρη ρωσική εκπαίδευση γλώσσα μιας ε, χώρας ε, μπορεί να πίσταται διακρίσεις. Δύσκολα όλα αυτά για τη Λετωνία, αλλά ε, στο μυαλό μας είναι η ασφαλής Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και σας εύχομαι καλή τύχη. Ο κύριος Μπαστινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητέ Πρωθυπουργέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ομιλία σας η οποία ήταν ρεαλιστική και εύρωστη αλλά και για τις ρεαλιστικές και συνεκτικές αξιολογήσεις και συνεισφορές σας. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπατε. Και εγώ και η χώρα μου, η Ρουμανία, βλέπουμε την Ρωσία όπως τη βλέπετε κι εσείς. Έτσι λοιπόν, πώς η Λετωνία αξιολόγησε την, ε, αξιολογεί την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και ποια θα πρέπει να είναι μελλοντική σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Άμυνας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ που παρουσιάζετε ένα όραμα εδώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ευχαριστώ και για τις παρατηρήσεις σας για την εσωτερική αγορά θα ήθελα να σας ζητήσω να διαβιβάσετε αυτό το μήνυμα στο Συμβούλιο, να πείτε ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα απειλούνται από την κομμουνιστική Κίνα. Αυτό που έχουμε τώρα ενωπιών μας και βλέπουμε είναι η ε, βιομηχανία των ευρωπαϊκών πλοίων που δέχονται επίθεση από τον κινέζικο ανταγωνισμό. Ε, βλέπουμε κάποια ναυπηγεία που πρέπει να πάρουν επιδοτήσεις ε, για να παροπλήσουν ε, τα παλιά πλοία τους και κατόπιν θα πρέπει να προσαρμοστούν ε, στις απαιτήσεις των κινέζικων εταιριών για την αυπήγηση των πλοίων. Πρόκειται για θέμη του ανταγωνισμό απέναντι στην ευρωπαϊκή, στον ευρωπαϊκό αυτοκλάδο. Και βλέπουμε ότι κατακτούν μια αγορά που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αγορά Ευρωπαίων ιδιωτών χωρίς να υπάρχουν κρατικές επιδοτήσεις. Όμως δεν θα πρέπει να είμαστε ανόητοι εδώ, θα πρέπει η Κομισιό να τα σκεφτεί όλα αυτά πολύ πιο ξεκάθαρα. Ο κύριος Ρανζέλ. Ευχαριστώ. Θέλω να σας συγχαρώ κύριε Πρωθυπουργέ για μία από τις πιο εμπνευσμένες ομιλίες που έχουμε ακούσει εδώ από πρωθυπουργούς. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για την πολιτική συνοχής και τα ταμεία συνοχής. Η Επιτροπή παρουσίασε μία πρόταση Όπου μια χώρα όπως η Λετωνία που έχει καταβάλει τόσες προσπάθειες και βρίσκεται σε χαμηλή θέση του χαμηλού μεσόρου χάνει 14% από το Ταμείο Συνοχής. Η Πορτογαλία χάνει 7%. Η Κροατία χάνει 5%. Είναι αποδεκτό οι πιο φτωχές χώρες να χάνουν κονδύλια από την πολιτική συνοχής. Πώς ο Πρωθυπουργό κάνει σκέφτεστε να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, ε, θα δράσει όπως η πορτογαλική κυβέρνηση που από ό,τι φαίνεται είναι πολύ ικανοποιημένη που η Κομισιόν από χώρε που είναι πιο φτωχέ από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Φιλανδία και έχουν σεβαστεί όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία να του αφαιρούνται κονδύλια από την πολιτική συνοχή. Ε, ποια μέτρα μπορούν και πρέπει να λάβουν οι χώρε αυτέ απέναντι στην πρόταση τη Κομισιόν. Ο κύριος Μίμικινς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, στην ομιλία σας δείξατε και το κινητό σας, μιλήσατε και για τον μύθο του Εσώπου. Οι διαφορές και η ποικιλομορφία στην Ευρώπη, ναι, υπάρχουν. Το γεγονός όμως ότι κάποιοι έστειλαν επιστολή στην λετονική κυβέρνηση για τον περιορισμό της εκπαίδευσης της γλώσσας των μενοτήτων τους αποκαλέσατε τρελούς. Ένας από αυτούς είμαι κι εγώ και οι συνάδελφοί μου, οι σοσιαλδημοκράτες. Η κυρία ε, Μάλλον είχατε και μια έκθεση πάρα πολύ καλή για το ξέπλυμα του χρήματος, αλλά δεν είπατε τίποτα για την ε, σύζυγό σας και για τις πωλήσει ακινήτων. Είπατε ότι είναι ο τύπος. Ναι, ίσως να μην είναι καλό ε, παράδειγμα. Αν θέλετε κύριε Κάνης να αλλάξετε την Ευρώπη, πρέπει να ξεκινήσετε από τον εαυτό σας. Δεν πρέπει να έχετε πια αμερικανική υπηκότητα. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάριντς. Θέλω να σας θυμίσω ένα πράγμα εγώ, κύριε Κάριντς. Πριν από 10 χρόνια θυμάμαι ότι πήγα στην ε, καντίνα και ήμουνα κάπως μόνος, γιατί και εσείς και κάποιοι συνάδελφοι με καλέσατε να έρθω και να μοιραστώ το γεύμα μου μαζί σας, να καθίσουμε μαζί. Δεν το ξεχνάω και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Και σας ευχαριστώ και για αυτά που είπατε χτες στην συνεδρίαση της ομάδας του ΕΛΚΑ. Τώρα, αναφερθήκατε όντως στο ξέπλυμα χρήματος και στην εγκληματικότητα. Και πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα στη χώρα σας. Και είπατε πώς ε, κυκλοφορούν εγκληματίες από τη μία χώρα στην άλλη. Εσείς τι θα θέλατε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία για να μειωθεί ακριβώς η νομοποίηση χρήματος από παράνομες ε, δραστηριότητες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι σας καλωσορίζουμε εσάς και τους συναδέλφους σας εδώ. Η κυρία Γκόμες. Σας ε, καλωσορίζω κύριε Πρωθυπουργέ. Ε, χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ και χάρηκα πάρα πολύ που συνεργαστήκα μαζί σας ε, στην ομάδα που διαπραγματεύτηκε την τέταρτη και την πέμπτη οδηγία για το ξέπημα βρώμικου χρήματος. Όπως και εσείς και εγώ έμαθα πάρα πολλά και λόγω των ε, επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα και για θέματα φορολογικά. Εκτιμώ αυτά που είπατε και σας στηρίζω ανεπιφύλακτα ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή κεντρική εποπτεία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και σας ερωτώ όμως, εσείς τώρα ως Πρωθυπουργός θα πιέσετε και για αυτά που έχουμε ζητήσει εμείς την πέμπτη οδηγία για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Επίσης για τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ ε, θα ασκήσετε εκεί πίεση γιατί βλέπουμε ότι διοχετεύονται πάρα πολλά χρήματα για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατικές οργανώσεις μέσα από το, τις απάτε απάτες ε, καρουσέλ. Και σα ερωτώ, θα πιέσετε για το MQV σε θέματα φορολογίας. Αυτό είναι καθοριστική σημασία ε, για να αντιμετωπιστεί κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το φορολογικό dumping το οποίο στρεβλώνει τους, ε, αγώνες θεμητού, τους κανόνες θεμητού ανταγωνισμού. Πρόεδρε, αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία στο Κοινοβούλιο και χαίρομαι πάρα πολύ που ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ε, βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Ε, Πρόεδρε, αυτά που είπατε σήμερα ήταν ε, ρεαλιστικά, θετικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί ο λαϊκισμός και ο εθνικισμός σε όλα τα κράτη-μέλη, από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Ο καλύτερος τρόπος είναι να καταδείξουμε ότι έχουμε ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν είναι μόνο μόνο ένα εγχείρημα ειρήνης, αλλά είναι και ένα εγχείρημα οικονομικής και κοινωνικής πρόοδου. Και το θεματολόγιο σας, Πρόεδρε, είναι σαφές. Θέλετε περισσότερο εμπόριο, να έρθουν οι φραγμοί που εμποδίζουν την κοινή αγορά, να μην υπάρχει προστατευτισμό σε περισσότερες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεμητός ανταγωνισμός. Αυτό είναι το θεματολόγιο που θα διασφαλίσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης, περισσότερες επενδύσεις, αλλά και περισσότερες ελπίδες για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί σας. Σας στηρίζουμε και εκτιμούμε όλα αυτά που κάνατε για τη δημοκρατία, την ελευθερία, για τις αξίες για τις οποίες τόσο εύγλωτα μιλήσατε σήμερα το πρωί. Ο κύριος Βάιντεν Όρτσερ δεν είναι εδώ. Μυρκούνεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε αντίθεση με άλλους συναδέρφους, ε, δεν είναι η τελευταία φορά που εγώ μιλάω εδώ στο ημικύκλιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάριν, τον Πρωθυπουργό, για την ενέργειά του, για την τόσο θετική ομιλία του για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα να συνεργαστώ μαζί σας αυτά τα χρόνια. Η προτεραιότητα ήταν η δημιουργία απασχόλησης επενδύσεων και εταιριών. Και πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Έχουμε περισσότερη απασχόληση στην Ευρώπη σήμερα, έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες επενδύσεις σε βαθμό όπως ήταν πριν από την κρίση. Όμω είναι δύσκολος ο διεθνή ανταγωνισμό, η ψηφιοποίηση αλλάζει τον κόσμο, οπότε εσείς τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνουν οι χώρε μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσουμε την οικονομία μας και την ανταγωνιστικότητά μας τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε κύριο Βαλσίτη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, Σήμερα θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την εξαιρετική ομιλία σας. Εσείς αναφερθήκατε στην ιστορία όχι μόνο της Λετωνίας, αλλά και των άλλων βαλτικών χωρών, της Εστονίας και της Λιθουανίας. Δεν θέλω να σας κάνω ερωτήσεις, αλλά βλέπετε είναι η τελευταία μου ομιλία στο ημικύκλιο αυτό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Και θέλω να κάνω έκκληση σε εσά, να σας ενθαρρύνω μια που είσαστε εκπρόσωπος του Συμβουλίου, να στηρίξετε την δημιουργία μιας αυθεντικής ενεργειακής αγοράς. Και δεύτερον, θέλω να κάνω έκκληση σε εσά να στηρίξετε επίσης και το πρόγραμμα για σιδηροδρόμους στην Βαλτική. Να επικεντρωθείτε επίσης σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και επίσης πολύ σωστά τίθεται και το θέμα των πληρωμών ε, γεωργικών κονδυλίων, κονδυλίων προς την γεωργία. Σας ευχαριστώ πολύ για ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε, κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κάραντς ε, γιατί στην ομιλία τον έφερε κάτι το πολύ σημαντικό, δηλαδή την ε, ψηφιακή εσωτερική αγορά. Και Κρίστιαν έχεις απόλυτα δίκιο ότι αν δεν ε, καταργήσουμε τους φραγμούς στην Ευρώπη, κυρίως την περιαγωγή, ποτέ δεν θα κατορθώσουμε αυτές τις πλατφόρμες που τους χρειαζόμαστε επιγόντως στην Ευρώπη, αυτές να είναι και αποτελεσματικές. Χρειαζόμαστε την δυνατότητα να μπορούμε να αγοράσουμε κάρτα SIM και στα 28 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χρειαζόμαστε ουσιαστικές εξελίξεις γιατί αυτές θα καθορίσουν τον ανταγωνισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που από κοινού εργάστηκαν για την κοινή αγορά και διασφαλίζουν τον μέλλον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Σας ευχαριστώ για αυτή τη φανταστική ευκαιρία Αγαπητοί συνάδελφοι, για πολλούς εδώ είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν ε, να μιλήσουν. Για μένα είναι πρώτη και τελευταία, καθώς πρόκειται για μένα. Είμαι ένα πολύ νέο μέλος, μόλις πριν 10 μέρες ε, ήλθα. Έτσι λοιπόν, για στατιστικούς λόγους, μήπως μπορείτε να σημειώσετε ότι είναι η πρώτη και η τελευταία μου παρέμβαση. Σας ευχαριστώ όμως ε, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα ήθελα να θέσω την ίδια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο Ρουμάνος συνάδελφος. Ποια είναι η άποψή σα για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Η Ρωσία έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, κατέχει, έχει κατα... παράνομα ε, μέρη της Ουκρανίας, τη Γεωργία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό και πώς ε, βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η δύσκολη σχέση με τη Ρωσία και ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα έπρεπε να σας δώσω και ένα δεύτερο λεπτό, αλλά δυστυχώς ε, δεν γίνεται. Συνάδελφος Αντρική είναι εδώ στην αίθουσα. Τότε ολοκληρώνεται το κατσιδιάι και θα δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό. Έχετε το λόγο, κύριε Κάρνης. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ κρατούσα σημειώσεις ε, όσο μιλούσατε. Έχω πάρα πολλές σημειώσεις ε, και φυσικά θα τις μελετήσω στο εγγύς μέλλον, τα θέματα. Συνοχή, γεωργία, μετανάστευση, νομιμοποίηση εισόδων, Κίνα, Ρωσία, άμυνα και τα λοιπά. Αν προσπαθούσα να απαντήσω, μάλλον θα μακρηγορούσα πολύ περισσότερο από ότι την πρώτη φορά, έτσι λοιπόν δεν θα το πράξω. Αλλά τι θέλω να κάνω, να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, ως πρώην ε, Ευρωβουλευτής θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την ευκαιρία, την ικανοποίηση και την τιμή που είχα να συνεργαστώ μαζί σας. Τα τελευταία δέκα χρόνια αλλά και η προηγούμενη θητεία ήταν ε, μια εξαιρετική εμπειρία για μένα. Από ό,τι φαίνεται συγκινούμε και κάπως. Όμως ε, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύ καλή συνεργασία. Πολλοί από εσά είπατε ότι πρόκειται για την τελευταία ομιλία σα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά εγώ μπορώ να πω ότι είναι η πρώτη μου ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω Πρωθυπουργό. Είμαι πολύ ικανοποιημένο λοιπόν γι' αυτό για να συνοψίσω τη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τέλεια, συνάδελφοι. Δεν είναι τέλεια. Και όταν οι ψηφοφόροι μας λένε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει να ακούσουμε τους ψηφοφόρους. Δεν πρέπει να λέμε όχι, όχι, όλα είναι τέλεια. Πρέπει να τους ακούσουμε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πραγματικέ ανησυχίε, είτε πρόκειται για τη δουλειά του, είτε πρόκειται για τη μετανάστευση, το κλίμα, την ασφάλεια. Αυτά τα θέματα είναι πραγματικά, αλλά επίσης έχουμε και πραγματικές απαντήσεις στα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε να εργαστούμε στο μέλλον ως ε, μια ένωση ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών ε, χωρίς να ε, δίνουμε ούτε ένα εκατοστό από την εθνική μας ταυτότητα ή της γλώσσας μας αλλά ε, θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Είμαστε μία Ευρώπη αξιών ελευθερίας, δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Ως λετονός μπορώ να πω ότι γνωρίζουμε τι σημαίνει να ζούμε ανελεύθεροι, χωρίς δημοκρατία και χωρίς κράτος δικαίου. Αυτό κανένας δεν χρειάζεται να το βιώσει ποτέ. έχουμε έναν βασικό τρόπο για να απελευθερώσουμε την οικονομική ανάπτυξη στην Οικονομική Ένωση. Και είναι κάτι απλό. Καλύτερη η αγορά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταλύσουμε τους φραγμούς της ενιαίας αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργήσουμε το περιβάλλον έτσι ώστε οι δικές μας εθνικές εταιρείες, οι ευρωπαϊκές εταιρείες να μπορούν να αναπτυχθούν και να είναι επιτυχείς παίκτες στη διεθνή σκηνή. Αυτό είναι στο χέρι μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο θέμα του μεταναστευτικού ενισχύοντας ε, τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό πρέπει να γίνει, γιατί όταν ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα μπορούμε να διατηρήσουμε ανοιχτά τα εσωτερικά σύνορα και να μην παρεμποδίσουμε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Μπορούμε να έχουμε μια ευφύ μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και πάλι το κλειδί είναι να διασφαλίσουμε ότι οι δυνάμεις της αγοράς υπάρχουν και λειτουργούν. Αφήστε την αγορά να απορριθμίσει τις ενέργειες και η πράσινη ενέργεια θα απογειωθεί, θα απογειωθούν οι ευφύς τεχνολογικές λύσεις, θα συμμετέχουν οι καταναλωτέ και η αγορά θα μα βοηθήσει να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Και σε ό,τι αφορά την κοινή μα ασφάλεια. Δεν βλέπω αντίφαση μεταξύ του να συμμετέχει κανείς στο ΝΑΤΟ όπως η χώρα μου και ισχυρότερη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέλος της ε, Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Δεν υπάρχει αντίφαση, αλλά θα πρέπει να πάμε ένα βήμα πιο πέρα από τη στρατιωτική ασφάλεια. Μιλάμε για την ε, ασφάλεια των πληροφοριών στο περιβάλλον πληροφοριών όπου ζουν οι πολίτες και θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά την εκπόνηση νομοθεσίας προκειμένου να δούμε ποια είναι η ευθύνη των πλατφορμών ε, κοινωνικής δικτύωσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ε, γιατί πολλές φορές η δράση τους παρεμποδίζει τη δημοκρατική ανάπτυξη. Συνάδελφοι, δεν χρειάζεται απαραίτητα να πολεμήσουμε τους λαϊκιστές. Οι πολίτες ακούν τους λαϊκιστές γιατί είναι δυσαρεστημένοι. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, βασικές αιτίε. Ως Ένωση είμαστε πιο ισχυροί, όπως το δεμάτι από τις βέργες. Παίρνεις μια βέργα και σπάει. Ένα, ένα έθνος μας μπορεί να σπάσει. Όλα τα έθνη παγκοσμίω είναι μικρά, αλλά ενωμένοι είμαστε σαν αυτό το δεμάτι από τι βέργε που δεν μπορεί να σπάσει και μπορούμε τη δική μα ιδέα του ελεύθερου αγοριού και του εμπορίου και του τρόπου ζωή μπορούμε να την προωθήσουμε στι άλλε αγορέ και όχι να αφήσουμε του άλλου να επιβληθούν σε εμά. Έτσι λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη που είναι της ε, αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, μαζί με τις αξίες της νέας αγοράς, να τις προωθήσουμε, να το κάνουμε αυτό με έναν ειρηνικό τρόπο, μέσω του διαλόγου, μέσω της συμμετοχής των πολιτών και έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά σας. Ευχαριστώ πολύ.